Dear colleagues, uh... καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε όλοι. Καλώς πρώτα απ' όλα τον Επίτροπο κύριο Γκίντερ Είναι παλιός γνώριμος εδώ στην Επιτροπή μας, τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εχθές συζητήσαμε την ασφάλεια ανεμφοδιασμού στο φυσικό αέριο. Δεύτερη προσέγγιση και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το 2010 ήταν η πρώτη δοκιμή, η πρώτη απόπειρα, <laughs> πάρα πολύ επιτυχημένη, ήταν δική σας πρωτοβουλία, εσείς εκπονήσατε την νομοθεσία, ε, πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα. Έχουμε επιτάπητος ε, πάρα πολύ συχνά τέτοια θέματα που ξεκίνησαν πριν από 5, 4, 3 χρόνια όταν είχατε εσείς το χαρτοφυλάκιο της ενέργειας. Τώρα είναι κάπως διαφορετικό το θέμα ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ κοντινό με το προηγούμενο και έχουμε ένα διαρθρωμένο διάλογο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανταλλαγή απόψεων λοιπόν το θέμα μας με τον κύριο Επίτροπο. Έχουμε ένα ψήφισμα για την ψηφιακή αγορά που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο στο Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια και πολλές προτάσεις απορρέουν. Θα συζητήσουμε, μάλλον στα εχθές συζητήσαμε το θέμα του ραδιοφάσματος. Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δέσμη της για την ψηφιοποίηση της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας μόλις αυτή την εβδομάδα. Ξέρουμε ότι σε λίγους μήνες έχουμε και άλλες προκλήσεις και άλλες προτάσεις ε, μπροστά μας και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ο διαρθρωμένος διάλογος βεβαίως είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα σας παρακαλούσαμε κύριε Επίτροπε να μας κάνετε μια ενημέρωση για το πώς προχωρεί η υλοποίηση του δικού σας προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 και να μας δώσετε και μία πρόγευση για το 2017. Πώς προτίθεται να κινηθείτε του χρόνου. Παρακαλώ κύριε Επιτροπέ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητέ καθηγητά Μπούζεκ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Στα πλαίσια της ψηφιακής μας πολιτικής, που έχει στόχο μια Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ένωση, φέτος έχουμε πάρα πολλά εγχειρήματα, νομοθεσία, ανακοινώσεις. Εγώ θα περιοριστώ σε πέντε κέντρα βάρους των εργασιών μας που έχουν σημασία και κυριαρχούν και στις δικές σας εργασίες της δικής σας σημαντικής επιτροπής. Πρώτον, αναθεώρηση των τηλεπικοινωνιών. Γενικά πολιτική στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Στο παρελθόν, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών είχε ως αντικείμενο τις τηλεπικοινωνίες και την τηλεφωνία. Υπήρξε ένας ξεχωριστός τομέας με δίκτυο δικό του, η κινητή τηλεφωνία με δεδομένα για επικοινωνίες, για συνομιλίες, για τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και για μεταφορά περιεχομένου. Ως εδώ. Σημαντικό μεν, αλλά ως εδώ. Τώρα όμως, όταν μιλούμε για νέες ψηφιακές υπηρεσίες, ο τομέας των τηλεπικοινωνιών καθίσταται πλέον εγκάρσιος, οριζόντιος, πέρα από την δική του ξεχωριστή ε, μεταφορά ε, έχει ε, να κάνει με αυτόματη οδήγηση, ε, με αυτόματη οδήγηση αυτόνομη, ηλεκτρική, μάλλον ηλεκτρονική ιατρική, τηλεϊατρική, αυτοκίνητα, ηλεκτρικά. Είναι το λεγόμενο διαδίκτυο των αντικειμένων, των Internet of Things. Άρα έχουν αυξηθεί και οι ε, υπηρεσίες που παρέχονται από την επικοινωνία κατακόρυφα και ε, η λέξη κλειδί είναι η σύνδεση. Οι ε, υποδομές, ευρυζωνικότητα, δορυφόρος, καλωδιακή και οι οπτικές είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι σημαντικότερες επενδύσεις των επομένων ετών. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει σε βάθος εξέταση και μελέτη έχουμε στόχους για διεύρυνση, για ανέβασμα και κατέβασμα, upload και download για την ευρυζωνικότητα στο δρόμο μέχρι το 2020. Για την επόμενη δεκαετία μέχρι το 2015 αυτό κυριαρχεί. και θα ε, γίνει ευρεία ε, διαβούλευση, αναλύσεις και θέλουμε μαζί σας και με τα κράτη-μέλη να έχουμε ένα σχέδιο ε, αξιόπιστο, σοβαρό για το πώς θα έχει η ψηφιακή υποδομή το 2025. Από τώρα θέλουμε αυτά να τα αποφασίσουμε. Μετά από διαβούλευση και επεξεργασία. Αν προσθέσουμε όλες τις ανάγκες για μεταφορά δεδομένων από τα social media, ε, ανέβασμα, κατέβασμα, streaming, από την κλασική τηλεφωνία, μέχρι ε, αυτό που χρειάζονται οι διάφορες πλατφόρμες ή διάφοροι κλάδοι της βιομηχανίας, 50 εκατομμύρια αυτοκίνητα και φορτηγά θα είναι συνδεδεμένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαστε 50 MHz ας πούμε, δεν πρόκειται για τέτοιες συχνότητες και δεν είναι ε, ο παράδεισος. Αυτά, πλέον συζητούμε για την κοινωνία των gigabyte και θα πρέπει με ευφυΐα ε, και με προσοχή να εργαστούμε έτσι ώστε οι επενδύσεις να γίνουν διασυνοριακά, πανευρωπαϊκά, ε, να φτάσουν σε όλη την επικράτεια και να πετύχουν. Η αναθεώρηση των τηλεπικοινωνιών είναι ένα και μόνο μέσο και εργαλείο προς την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευφύης, έξυπνες προϋποθέσεις και το πλαίσιο εκείνο έτσι ώστε να υποστηριχθεί η, ε, επικοινωνία, η τηλεπικοινωνία και ο κλάδος από οικονομική υποστήριξη για να μπορεί να ε, κάνει τις σωστές επενδύσεις. Δεύτερον, η πολιτική του ραδιοφάσματος για τις συχνότητες. Θα πρέπει μέχρι τώρα να υπάρχει καλύτερος συντονισμός και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το καιρό και σας ευχαριστώ συζητάτε το θέμα αυτό και με ένταση εργασίας. Είναι η πρώτη νομοθεσία μας για ε, ε, το ζήτημα των 500 MHz. 700, συγγνώμη. Αυτό ήταν και ένα αποτέλεσμα των εργασιών του Πασκάλ Λαμή. Χρειαζόμαστε ένα νέο κανονισμό για ε, τη ζώνη του ραδιοφάσματος στα MHz μεταξύ διαφόρων χρηστών. Πώς θα τα μοιράζονται ε, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες. Και αν έρθει το 5G, η πέμπτη γενεά ε, κινητής τηλεφωνίας, τότε η ζώνη των 700 MHz χρειάζεται συντονισμό για τη χρήση. Και ερχόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Η Renault, η Mercedes-Benz, τα νέα αυτοκίνητα ε, της κατηγορίας ε, η BMW, όλες οι βιομηχανίες χρειάζονται υποστήριξη και έχουν και όλους τους προμηθευτές ε, που εργάζονται για τις εταιρείες αυτές και από το 2020 θα καταστήσουν δυνατό το αυτοκίνητο που θα κυκλοφορεί χωρίς οδηγό. Τα αυτοκίνητα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει διασύνδεση, ε, το διαδίκτυο που χρειάζεται για να κυκλοφορούν αυτά τα αυτοκίνητα. Θα πρέπει λοιπόν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι η Acer, η OEM, ε, οι κατασκευαστές γιοταχή και φορτηγών και από τη μια και από την άλλη ε, η τηλεπικοινωνία γιατί ταυτόχρονα θα πρέπει να συζητήσουν όλοι αυτοί για να συντονιστούν. Η αγορά θα έχει καλά αυτοκίνητα, αλλά θα μπορούν και να κυκλοφορούν με αισθητήρε στα αυτοκίνητα, με ψηφιακά στοιχεία στα αυτοκίνητα και θα πρέπει η τηλεπικοινωνία να τους δίνει τη δυνατότητα να μεταδίδονται και να μεταφέρονται αυτά τα δεδομένα και όχι σε ένα κάποιο αυτοκινητόδρομο για λόγους δοκιμής του αυτοκινήτου, όχι, παντού και στο μέλλον Αδρυμό και στην Ήπεθρο και σε κάθε χωριό ας πούμε και διασυνοριακά. Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι ε, τα σύνορα δεν τα βλέπετε στην Ευρώπη από τα νομίσματα ε, γιατί έχουμε νέο νόμισμα ε, ούτε από τον έλεγχο στα σύνορα που δεν υπάρχει και ελπίζω και στον Μπρένερ να μην υπάρχει αυτό αλλά το βλέπετε γιατί

Θα πρέπει η πολιτική ραδιοφάσματος λοιπόν να συντονιστεί πανευρωπαϊκά και να υπάρχει κάλυψη σε όλη την επικράτεια ψηφιακή στη γενιά των 5G πλέον. Και 5G ε, PPP προχωρεί. Ε, γίνονται διάφορες συμφωνίες, συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Συνεργασίες με τρίτες χώρες, με την Νότια Κορέα, φιλοδοξεί η Ευρώπη να είναι εκείνη η επικράτεια που να υπάρχει βάση ε, για σωστή λειτουργία του 5G και να μπορούν να παρέχονται όλες αυτές οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Όλα αυτά αφορούν τις τηλεπικοινωνίες και την αναθεώρηση που θα έχει κατά τη διάρκεια του 2016. Διότι α, στις εργασίες μας, και θέλω να το συμπληρώσω αυτό, είναι το θέμα του Μπερέκ. Γνωρίζετε εσείς το φορέα αυτό στην Επιτροπή σας και γνωρίζετε και το Acer. Το Κοινοβούλιο γνωρίζει και άλλα δίκτυα ρυθμιστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράδειγμα, ε, υποπτία των ασφαλίσεων, υποπτία των τραπεζών. Ε, γενικά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του τομέα αυτού. Έχουμε εθνικές ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, οι κεντρικές τράπεζες, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία εποπτεύει. Και στην ενέργεια έχουμε το Acer που παγκοσμίως μάλλον ε, γενικά έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από τον BEREC. Σήμερα θα, θα συναντηθώ με τους ρυθμιστές του Μπέρεκ, που είναι πολύ ισχυροί οργανισμοί ρυθμιστικές αρχές επιτόπου. Αλλά γενικά ε, χρειάζεται να γίνει μια στρογγυλή τράπεζα, ένα ε, think tank, μια ομίγυρη, ένας γενικός ε, καφές ας πούμε για να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Και για να τα πω πάρα πολύ ειλικρινά τα πράγματα, εάν σήμερα η Ευρώπη γνώριζε την πρώτη μέρα της δημιουργίας, εγώ θα δημιουργούσα και θα πρότεινα μία ρυθμιστική αρχή για όλα. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε 28 και έχουμε και την Νορβηγία, την Ελβετία, τα Δυτικά Βαλκάνια, τους εταίρους μας που συμμετέχουν. Αλλά θέλω να τους βλέπω αυτούς πιο συχνά στην στρογγυλή στράπεζα του Μπέρεκ, που είναι οι διευθυντές των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών και να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες. Οι ρυθμιστές των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιών είναι αυτοί. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο σημείο που σας ανέφερα για τις τηλεπικοινωνίες. Δεύτερον, όπως είπατε, την Τρίτη παρουσιάσαμε τη δέσμη μας για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, μου έκανε εντύπωση ότι στην ψηφιακή οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δραστηριοποιείται πάρα πολύ, αλλά το θέμα μιας ε, ψηφιακής βιομηχανικής πολιτικής, δηλαδή πώς μπορούμε τις εταιρείες μας και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες να τις βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, τις θέσεις εργασίας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή επανάσταση ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τώρα αυτό απουσίαζε από το πρόγραμμα και το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα έχουμε εκπονήσει ένα ευρύτατο πακέτο, μία δέσμη ολόκληρη, που πέρυσι παρουσιάσαμε στο, και ανακοινώσαμε στο Ανόβερο που είναι η παγκόσμια έκθεση ε, και τη Δευτέρα έχουμε μια διάσκεψη και πάλι στην Τσέμπιτ που είναι η έκθεση ε, βιομηχανίας στο Βούργο, στο Ανόβερο συγγνώμη. Και θέλω ε, πραγματικά να επικεντρωθούμε σε αυτή την προσπάθεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, είναι τέρος. Ε, θα έρθει ο Ομπάμα, θα έρθει και η μισή του κυβέρνηση, θα έρθουν πολλοί διευθυντέ και στελέχοι επιχειρήσεων και ε, ε, διευθυντές, αλλά πολύ περισσότεροι από την ψηφιακή οικονομία, από τη Microsoft. Οι Αμερικανοί έχουν άλλη προσέγγιση, έχουν το big data, ε, κυριαρχούν στα ψηφιακά, έχουν πλατφόρμες με πολύ μεγάλη οικονομική υποστήριξη και θέλουν να ανακτήσουν, δηλαδή είναι η ηγετική δύναμη ε, σε αυτά τα θέματα, αλλά όχι ε, στην βιομηχανία. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε, ας πούμε, οργανώνουν τη διασύνδεση, η Ρενό, η BMW φτιάχνουν τα αυτοκίνητα και θα πρέπει όλοι αυτοί να συνεργαστούν για να φτάσουν στον πελάτη. Και εμείς θέλουμε να αντισταθούμε σε αυτό και να ε, κάνουμε μια ευρωπαϊκή προσπάθεια με κάθε φιλία, γιατί είναι εταίρος μας οι ΗΠΑ. Σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν δίκτυα ε, το καταπούλτο ε, στις, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις κατοχώρες Smart Factory, στη Γαλλία Industry Industrie du Futur, στη Γερμανία Βιομηχανία 4.0 και στην Αυστρία αντίστοιχα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο δικτύων στην Ευρώπη και να ελέγξουμε πού η συνεργασία βοηθάει ή πού σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγαλύτερο νόημα να συντονιστούμε παρά να έχουμε 28 παράλληλα ασύνδετα δίκτυα στα κράτη-μέλη. Η τυποποίηση είναι πολύ σημαντική εδώ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέλουμε να προωθήσουμε την τυποποίηση. Έχουμε εντοπίσει τους τομείς στο IoT, στην ασφάλεια, στο διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο, το 5G όπως σας είπα. Ε, η τυποποίηση επίσης των clouds, των ηλεκτρονικών ε, νεφών και θέλουμε τα αρμόδια ιδρύματα και οργανισμοί τυποποίησης να εξυγχρονιστούν, αν χρειαστεί και με νομοθεσία, για να προχωρούν ε, σε τυποποίηση ευρωπαϊκή. Μόνο έτσι θα μπορέσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα να γίνουν και παγκόσμια. Αλλιώς δεν πρόκειται να πετύχει η προσπάθεια αυτή. Επίσης, υπάρχουν μερικά μεγάλα έργα που πρέπει να προωθηθούν πανευρωπαϊκά. 5G με 700 εκατομμύρια από το προπολογισμό μας, το ανέφερα. Αναφέρω και το θέμα των super υπολογιστών, high performance, υψηλής απόδοσης, στη δεκαετία του 80. Οι έξι μεγαλύτεροι υπολογιστές του κόσμου ήταν στην Ευρώπη. Σήμερα είναι δύο και σε σελίδα ε, ε, στην ε, ένατη θέση είναι στη Γερμανία και στην 8η ε, ε, ένας υπολογιστής στη Ζηρίχη. Οι 6 στους 10 μεγάλους βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα και στην Νότια Κορέα είναι γιγαντιές. Γι' αυτό στο σχέδιο Juncker ζητούμε συγχρηματοδότηση και δίνουμε κίνητρα από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό με προκηρύξεις διαγωνισμών. Είμαστε επαφή με διάφορους ομίλους δεν θα έχουμε φυσικά 28 υπερυπολογιστέ, αλλά με ομιλού στη Γερμανία, ε, από τη Στουτγάρδη, στο Λουξεμβούργο ή αλλού και στην ε, Γαλλία, στην Ιταλία. Τρει, τέσσερι, πέντε από του δέκα καλύτερου, μεγαλύτερου υπολογιστέ στον κόσμο θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Αλλά να έχουν πρόσβαση ε, όλοι οι Ευρωπαίοι, είτε είναι ερευνητέ, είτε είναι οικονομία και διάφοροι φορεί που χρειάζονται τα στοιχεία αυτά για τη δουλειά του. Θέλουμε να έχουμε ένα ερευνητικό cloud. Η ψηφιοποίηση λοιπόν της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ένα πακέτο το οποίο καταθέσαμε την ε, Τρίτη και τις επόμενες εβδομάδες είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι συζητήσεις θέλετε. Τρίτη ε, προτεραιότητα, η ασφάλεια στο διαδίκτυο και στον κυβερνοχώρο. όπως και στην έκθεση Τσέμπιτ του ε, Νοβέρου, όπως και στην άλλη παγκόσμια διάσκεψη, ήταν δύο τα θέματα, το 5G και η ασφάλεια του δικτύου. Ε, ε, βιομηχανική κατασκοπία, τρομοκρατία, χακάρισμα, ένα σωρό απειλές έχουμε στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Θα πρέπει να προστατεύεται η οικονομία μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ε, ναι, ευρωπαϊκή υπόθεση αυτή ασφάλεια στον κυβερνοχώρο επίσης, ΖΙΤ που θα ξεκινήσει ε, το καλοκαίρι με μέσα από το ορίζον 2020 θα χρησιμοποιηθούν κονδύλια για συγκεκριμένα έργα, αλλά ήδη σας εξαγγέλω ότι η επόμενη οδηγία δεν θα είναι η τελευταία. Σε ένα με ενάμιση χρόνο μέσα θέλω με συμμετοχή της ΕΝΙΖΑ ε, αλλά και των Εθνικών Αρχών ε, Ασφάλειας και με όλους τους Ενδεχομένω φορεί θέλω διεύρυνση και εμβάθυνση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και της ευρωπαϊκής κουλτούρας και νοοτροπίας για την ασφάλεια και προστασία από το ηλεκτρονικό έγκλημα. Με επιστοποιήσεις, με επισημάνσεις, με φορείς που θα κάνουν διάφορους ελέγχους. Τέταρτο σημείο από τα πέντε είναι οι πλατφόρμες επιγραμμικές. Εδώ τίθεται το εξή βασικό ερώτημα. Τι γίνεται με τις πλατφόρμες αυτές. Χρειάζεται ρύθμιση ο κλάδος. Copyright. Κάνουμε μεταρρυθμίσεις στις νομοθεσίες και πλατφόρμες online. Ε, ε, οπτικοακουστικά και αντίστοιχη οδηγία. Και ε, εκτός από τα κανάλια και το Spotify και το Amazon, υπάρχει το YouTube, υπάρχουν νέοι πάροχοι για εικόνες που δεν ε, ε, υποχρεώνονται ε, να προστατεύουν τους ανηλίκους. Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν εκεί. Λοιπόν, τι γίνεται με την υπόθεση του ανταγωνισμού, του θεμητού ανταγωνισμού. Χρειάζεται συμπλήρωση αυτή η κατάσταση που ήδη υφίσταται και μια πλαισίωση. Και πέρα από ε, τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright και την αναθεώρηση των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο χρειάζεται γενικά να εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές και νομικά δεσμευτικές. Ε, γίνεται η διαβούλευση που τελειώνει και το ε, φθινόπωρο θα έρθει πρόταση. Πέμπτο, προστασία των δεδομένων. Την περασμένη εβδομάδα το Κοινοβούλιο ενέκρινε και την οδηγία και το βασικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων για να υπάρχει ένας βασικός κανονισμός στην Ευρώπη και τώρα η οδηγία για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες ε, χρειάζεται αναθεώρηση ή privacy λέγεται αυτό, ιδιωτικότητα ή ιδιωτική ζωή ε, ε, στον ηλεκτρονικό κόσμο. Αυτά είναι τα πέντε βασικότερα, δεν είναι όλα, δεν είναι εξαντλητικός ο κατάλογος ε, και είναι θέματα για τα οποία είστε εσείς αρμόδιοι επί της ουσίας στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Μιλήσατε για πάρα πολλά πράγματα, για την ψηφιακή αγορά, για τις επικραμμικές πλατφόρμες και ούτω καθεξή. Τώρα περνάμε στη συζήτηση. Εξ ονόματος πολιτικών ομάδων έχετε δύο λεπτά. Οι συντονιστές και ένα λεπτό οι βουλευτές. Θα τελειώσουμε έτσι 10 και 10. Καταλάβετε παρακαλώ ότι δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Δύο λεπτά, δεκαστήριο Βέρα. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ Επίτροπε. Επειδή είστε σήμερα εδώ μαζί μας, είμαστε σε κρίσιμη φάση. Σύντομα θα, έχουμε, είμαστε στο ίμιση αυτής της θητείας. Είπατε ότι το αριθμιστικό πλαίσιο για την ηλεκτρονικέ επικοινωνίε είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την ε, μεταμόρφωση της ψηφιακή ενιαία αγοράς. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως τελικά οι τηλεπικοινωνίες είναι ένα είδος, ε, μάλλον παρέχουν ε, τη σπονδυλική στήλη για τα ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Είναι λοιπόν καιρός να τελειοποιήσουμε αυτό το πολύτιμο μέσο. Το τελευταίο ήταν το 2009. Εφτά χρόνια έχουν περάσει. Αυτό είναι μια αιωνιότητα για τον ψηφιακό τομέα. Θέλω να αναφέρω τρεις κατευθύνσεις γραμμέ που κατά τη γνώμη μου πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχάς, πιο απλή και αναλογική ε, ε, ρύθμιση, έπειτα ε, ρυθμιστική συνέπεια λόγω των αλλαγών, λόγω των νέων υπηρεσιών, και δίκαιος συντονισμός για τη διαχείριση του φάσματος, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις που απαιτούν, μάλλον, μια ανάμεκτη προσέγγιση, δηλαδή αποκλειστικές άδειες, ε, ε, γεωγραφική ε, κατανομή και ούτω καθεξής και πολλά άλλα που οι προηγούμενες που θα οδηγήσουν σε καλύτερο συντονισμό των συχνοτήτων. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές νομίζω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην αναθεώρηση. Νομίζω πως συμφωνούμε μαζί σας και πιστεύω πως είστε στο σωστό δρόμο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μίκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, περιστατωμένη σας εισήγηση. Είναι η πρώτη φορά που ακούω έναν επίτροπο να μας παρουσιάζει μία τόσο ευρεία εικόνα και οπτική και όραμα για αυτόν τον τομέα των επικοινωνιών και της ψηφιακής ε, αγοράς. Έχω ερωτήσεις. Σε συμφωνώ με αυτά που είπατε ότι χρειάζεται μια εφαρμοστική αρχή και εκτελεστική αρχή. Πρέπει να αποφύγουμε τις ε, παρακάμψεις της αγοράς ε, με υπερβολική νομοθεσία. Ίσως και σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να απορριθμιστούν τα πράγματα, όμως ε, πρέπει να δούμε όλες τις όψεις του νομίσματος. Όσον αφορά το, το σύστημα του cloud, αυτά τα στοιχεία που τοποθετούνται. Πρόκειται ας πούμε για προσωπικά ιατρικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών. Θα βρίσκονται εδώ ή θα είναι εκτός της Ένωσης, που αποθηκεύονται και αν είναι εκτός ποιος θα ελέγχει αυτά τα στοιχεία. Κάτι ακόμα, όλα τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούν εφαρμογές. Ακόμα και για να στείλει ένα mail κανείς, χρειάζεται μια ε, εφαρμογή. Δηλαδή μπορεί κανείς να έχει ε, ένα σωρό προσωπικά στοιχεία. Έχουμε έναν κατάλογο επαφών, ας πούμε, όταν υπάρχουν επαφές ακόμα και οικονομικού χαρακτήρα. Ε, τι γίνεται με όλα αυτά. Δεν μπορούμε δηλαδή να κρύψουμε τίποτα ούτε καν σε ένα προσάρτημα, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι στη διάθεση όλων και αυτό είναι παράδεκτο. Σας ρωτώ λοιπόν, τι σκοπεύετε να κάνετε, θα φτιάξετε κάποια οδηγία, τι θα κάνετε για να γνωρίζετε ποιες είναι οι παράμετροι που μπορούν να είναι γνωστές στην Ευρώπη και τι, τι έχετε σκεφτεί γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σας. Είναι καλή αυτή η παράδοση και την αξιολογούμε. Για το πρόγραμμα δράση που αποφασίσετε, έχω μια ερώτηση για το cloud computing. Το υπολογιστικό νέφος είναι σημαντική υπόθεση και να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό cloud για την έρευνα, την οικονομία και τα πανεπιστήμια. Είναι καλή αρχή, μήπως θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω. Και συζητήσαμε για τα ευρωπαϊκά cloud για τα πάντα. Ε, γιατί όλοι έχουμε το ίδιο πρόβλημα ω πολίτε αυτή την Ένωση Υπάρχει μαζική παρακολούθηση από την NSA που εξακολουθεί. Ε, προτίθεται να κάνετε τίποτα παραπάνω ή είναι μόνο για τα πανεπιστήμια, την έρευνα και την οικονομία. Δεύτερη ερώτηση. Κέντρα αριστείας για τις τεχνολογίες του διαδικτύου. Μπορείτε να επεκταθείτε αυτό πώς θα λειτουργήσει και θα υπάρξει και ένα θεματολόγιο για επαγγελματικά προσόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και τελευταία ερώτηση, η οδηγία για το e-privacy αναθεωρείται και αλλάζει για την ε, ιδιωτική ζωή στον κυβερνοχώρο. Ε, ξέρετε ότι κατέρευσε και απερίφθη η οδηγία για την προληπτική αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Στην παρούσα οδηγία αυτό θα επανέλθει ή δεν θα παίξει κανένα ρόλο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κάλλας. Danke. Danke, Herr Kommissar, dass Sie hier kommen und Rede und Antwort stehen. ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα άκουσα για τη τεχνολογία εχμής και πώς θα προχωρήσουμε. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, πολύ σημαντικά και πολύ καλά τι μέτρα έχουν ληφθεί έτσι ώστε ε, από την τεχνολογία εχμής να μπορέσουν όλα αυτά να φτάσουν ε, προς τα κάτω στις μικρές επιχειρήσεις, στις μεσαίες επιχειρήσεις, να ξεφύγουμε από την τεχνολογία εχμής και τη, τη μεγάλη στην Ευρώπη, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και με τους μικρούς. Και έχω και μια ερώτηση για τη διαφάνεια. Πριν από λίγες μέρες ήρθατε στην Αυστρία σε μια συνάντηση υψηλού επίπεδου με ε, εκπροσώπους λόμπι. Όταν υπάρχει τέτοια υψηλή εκπροσώπηση, αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνονται πιο διαφανώς, ε, να τα ξέρουν οι πολίτες, να τα ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι, η κοινή γνώμη, δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά στις Βρυξέλλες, να έχουμε και εμείς πρόσβαση. Μπορείτε να μας πείτε λίγο τι σας είπαν εκεί οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των εταιρεών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορέλη, ευθυντή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, που είστε εδώ. Εσείς σωστά εκφράσατε τις προτεραιότητες της Κομισιόν όσον αφορά την ψηφιοποίηση της ε, βιομηχανίας. Όμως δεν μιλήσατε για χρονικά όρια. Δηλαδή θα ήθελα να γνωρίζω πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να υλοποιήσετε αυτέ τις προτεραιότητε και πάντοτε σε σχέση με χρονικά περιθώρια. Εχθέ μιλήσαμε για την πολιτική του φάσματος σε αυτήν την Επιτροπή και ορισμένοι συνάδελφοι εξέφρασαν την βούληση για ε, ευελιξία όσον αφορά το φάσμα. Εγώ και η ομάδα μου ωστόσο είμαστε αρκετά αυστηροί γιατί πιστεύουμε ότι η τεχνολογία τρέχει πολύ γρήγορα ήδη τα, οι προθεσμίες που μας υποδείξατε είναι πολύ ε, μακριά. Είστε έτοιμοι να σεβαστείτε αυτές τις προθεσμίες και ενδεχομένως και να τις ε, φέρετε και πιο κοντά, να τις ε, μικρύνετε. Ευχαριστώ. Σαφχόζερ. Ευχαριστώ. Λυπούμε που έφτασα καθυστερημένα και που δεν μπόρεσα να είμαι εδώ και χτες για οικογενειακούς λόγους. Έχω παρατηρήσεις επί της ουσίας σε σχέση με την κυριαρχία και την ε, αντοχή. μιλάτε για 12 μεγάλους σερβερ, δύο είναι ε, στη Σκωτία και στη Μεγάλη Βετανία. Τι πιστεύετε όσον αφορά την αντοχή του ίντερνετ και της υπηρεσίας για τη δημιουργία ενός μεγάλου σερβερ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή ευρωπαϊκό επίπεδο στο κέντρο της Ευρώπης. Δεύτερον, τι γίνεται με τα λογισμικά. Έχετε σε επίπεδο λογισμικών και ε, υπαλλήλων μια στρατηγική, ευρωπαϊκή στρατηγική κυριαρχίας ε, δηλαδή ε, μηχανές ε, αναζήτησης, Google, Facebook, πλατφόρμες ανταλλαγών. Οι Ρώσοι έχουν φτιάξει ένα ανεξάρτητο σύστημα, οι Κινέζοι επίσης. Η Ευρώπη έχει κάποια στρατηγική ανεξαρτησίας η παρατήρησή μου αφορά και την αντοχή. Καλύτερη, ο καλύτερος τρόπος να καταστήσουμε αυτό το σύστημα ανθεκτικό δεν είναι να επιμείνουμε στα κράτη και την αλληλοσύνδεσή τους. Εμείς είμαστε υπέρ της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε ανθεκτικό το σύστημα και το cloud επίση είναι να έχουμε μια εθνική στρατηγική έκαστο και στη συνέχεια μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα διευκολύνει τι ανταλλαγέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πράγμα που θα μα δίνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αν ένα σύστημα δηλαδή καταρρεύσει, να έχουμε διαφορετικέ εναλλακτικέ διαθέσιμε. Γι' αυτά θα, τις τρεις παρατηρήσεις ήθελα να σας ρωτήσω και ε, αυτές αφορούν ε, βεβαίως την κυριαρχία σας. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε ένα μακρύ κατάλογο μονόλεπτων ε, παρεμβάσεων. Μπόνι, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, περιστατωμένη σας εισήγηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε πως η ψηφιακή επανάσταση αποτελεί ε, μεγάλο μοχλό αλλαγής για την οικονομία μας και την κοινωνία μας. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα καλύτερο ρυθμιστικό και μη ρυθμιστικό πλαίσιο. Όταν μιλάμε για τις υποδομές είναι σαφές ότι ο στόχος είναι η πέμπτη γενεά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν, θα να είμαστε προσανατολισμένοι στις επενδύσεις, στην ισορροπία, στον ανταγωνισμό. Όλα αυτά πρέπει να συμβαδίσουν και επίσης χρειάζεται συντονισμός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα και τα αυτόνομα αυτοκίνητα άνευ οδηγών, να, είναι, να αποτελέσουν την δυνατότητα για καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τις ε, εθνικές οργανώσεις. Η δήλωση του Άμστερνταμ με αυτού ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση γιατί μιλάμε εδώ για σε αυτή τη δήλωση για την ανάγκη νέων στάνταρ. Εάν θέλουμε διασυνδεσιμότητα, σας ευχαριστώ πολύ Μπλανκο Λόπες, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την εισήγηση και για το μεγάλο και φιλόδοξο πακέτο που μας παρουσιάσατε αυτή τη βδομάδα. Με αυτό θέλετε να κινητοποιήσετε 50 εκατομμύρια ευρώ ε, επενδύσεις σωστές, ε, ε με συγχωρείτε, Μιλάτε λοιπόν για 50 ευρώ, 50 ε, εκατομμύρια ευρώ. 500. 500, 500 εκατομμύρια τα οποία θα είναι ε, προσανατολισμένα σε αυτό το φιλόδοξο πακέτο. Επίσης μας μιλάτε για το ότι θα δημιουργηθούν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μέχρι το 2020 και ιδιαίτερα στον τομέα της ρομποτικής. Θέλετε να προωθήσετε την, ε, τον προσανατολισμό των εργαζομένων προς αυτούς τους τομείς. Όμως βλέπουμε ότι η στρατηγική που μας ε, παρουσιάζεται σε αυτό το τομέα δεν παρουσιάζεται αρκετά λεπτομερώς όσον αφορά τους κοινωνικούς φορείς και τον ε, κλάδο. Επίσης, τις τελευταίες μέρες, ευχαριστώ πολύ, έχουμε... Είδαμε το σκάνδαλο Woodbook στην Αμερική. Τι είναι, ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτρο Πέτσεγκερ για τις ε, πολύ καλές και σημαντικές ε, παρατηρήσεις σας για τη ψηφιοποίηση της ε, βιομηχανίας. Σημαντική βάση είναι και οι υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Το είπατε και χθες ξεκάθαρα στη συνέντευξη τύπου ότι θέλουμε να θέσουμε τα θεμέλια για μια κοινωνία gigabyte η Internet Economy Foundation έβγαλε μια μελέτη πάρα πολύ σημαντική που λέει ήδη το 2025 τα τρία τέταρτα των γερμανικών νοικοκυριών θα χρειάζονται ε, ευρυζωνικό δίκτυο το οποίο ε, δεν καλύπτεται από τη σημερινή τεχνολογία. Και θα πρέπει να αποφασίσει ο αρμόδιος φορέας τι θα κάνει ε, και πώς θα προχωρήσει με την τεχνολογία vectoring. για να υπάρχει υποδομή εχμής ε, στην Ευρώπη, αλλά ακόμα δεν βρισκόμαστε εκεί. Για ψηφιοποίηση της οικονομίας και της βιομηχανίας χρειαζόμαστε θεμικό, ε, ε, θεμητό συγγνώμη, ανταγωνισμό και οπτικές ίνες στην τεχνολογία και στις υποδομές μας. Πώς το βλέπετε. Για τη Γερμανία ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι. Ευχαριστώ. Ο κύριος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πώς συνεργάζεται με το ITU της Γενέβης και τι γίνεται με τη διεθνή περιαγωγή. Υπάρχει τώρα μια σύσταση για cost-based roaming, περιαγωγή με βάση το κόστος. 2 με 3 ευρώ κάνει ένα gigabyte στη χώρα μας, αλλά αλλού μπορεί να κοστίζει μέχρι και 19.000 ευρώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτίθεται στο 5G ε, να συνεργαστεί με τον αρμόδιο φορέα στη Γενέβη για να μην καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 40% των Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν ε, καθόλου ή έχουν ελλειπείς ε, ψηφιακές δεξιότητες. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιγόντως σχετική κατάρτιση για επιτρέψουμε και στους νέους ε, να μπουν ε, με ύψηλες δεξιότητες στην αγορά εργασίας ε, στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, να προωθήσουμε τις θετικές επιχειρήσεις και να επιτρέψουμε σε όλους τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υγεία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν. Πρέπει λοιπόν να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα στις επιμέρους κοινότητες και μέσα στον Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να αφορά τους ανθρώπους, ποιοτικές θέσεις εργασίας και οικονομική μεγέθυνση για όλους τους πολίτες πολίτες και όχι μόνο για ορισμένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίβλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, για ε, ε, τις παρατηρήσει σα πάντα είναι χρήσιμο και εμπλουτιστικό να συζητάει κανεί μαζί σας. Μιλήσατε για την ε, διασύνδεση, το connectivity, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν εκεί υποδομές, συμφωνούν όλοι. Πριν από τρει εβδομάδες είχε έρθει εδώ στην Επιτροπή μας ο κύριος Μόλτερερ, επικεφαλής του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, που μας είπε ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να χρηματοδοτηθούν ε, ψηφιακές υποδομές. Αλλά προς το παρόν είναι περιφερειακή και περιθωριακή συμμετοχή του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων είναι μόλις της τάξης του 7%. Θα πρέπει πανευρωπαϊκά λοιπόν να γίνει αυτή η προσπάθεια και στη ρύθμιση δεν ξέρω χρειάζονται κάποιες αλλαγές είμαι σε κάποια σύγχυση. Κάναμε τόσο πολλά το Connecting Europe Facility. Καλά, έχει χάσει κάποια χρήματα η διευκόλυνση αυτή. Έχουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, αλλά δεν βλέπω και καμία τεράστια πρόοδο. Έχετε άλλε ιδέε. Δεύτερον, τα μεγάλα έργα. Στα πλαίσια τη ψηφιοποίηση ε, τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία, Μπορείτε να μας δώσετε μερικά παραδείγματα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε αυτή τη φάση όπου προσπαθούμε να προστατεύουμε κόσμο ε, ε, ενώ πολλές χώρες ορθώνουν σύνορα στον κόσμο που έρχεται, το τομέα το ψηφιακό, τα σύνορα έχουν ε, καταργηθεί. Και θέλω να θέσω τι εξής ερώτηση. Εγώ είμαι εισηγητή αυτή τη Επιτροπή για τον κανονισμό που στόχο έχει να εξασφαλίσει τη δυνατότητα μεταφοράς των υπηρεσιών διασυνοριακά. Είναι μια πρόταση τη Κομισιόν που είναι απλή ε, και σαφή. Δύο όμως κρίσιμα σημεία περιλαμβάνει. Πώς ορίζουμε την κατοικία του καταναλωτή, πώς ορίζεται και το άλλο είναι ποια είναι τα κριτήρια για να εγκρίνουμε τη συνελόγω υπηρεσία. Πώς μπορούμε να διευκρινίσουμε αυτές τις καταστάσεις χωρίς να υπάρξει έλλειμμα δημοκρατικό και έπειτα ε, το κίνδυνο στην ενιαία χώρα είναι η συγκέντρωση των ε, φορέων σε ισχυρότερε ε, αγορές, οι περιφέρειες της αγοράς εις βάρος των πιο αδυνάμων περιφερειών. Ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ και Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω μερικές παρατηρήσεις. Ε, σωστά είπε ο Επίτροπος ότι χρειαζόμαστε 100% ε, κάλυψη στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια για το διαδικτύο. Αυτό δεν υπάρχει ούτε καν στους ε, αυτοκινητοδρόμους ούτε στην Τσεχία. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στην ηλεκτρονική κλίση από τα αυτοκίνητα. Το λεγόμενο e-call είναι σημαντικό για την ασφάλεια. Αν ε, πάτε στην Ιαπωνία ή στην Νότια Κορέα, ε, δεν έχετε δυνατότητα, δεν λειτουργεί το κινητό εκεί. Πρέπει να τυποποιήσουμε κάπως και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, θα πρέπει να περάσουμε όντως στην ψηφιακή εποχή και είναι πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την κοινωνική διάσταση. Στην Τσεχική Δημοκρατία το 2011 περάσαμε στο ψηφιακό σήμα, κάναμε αυτή τη μετάφαση, τώρα θα έρθει για δεύτερη φορά. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά όμως για να τα υποστηρίξει όλα αυτά. Ο κύριος Έλλερ, ε, σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε σε αυτά τα θέματα και που ε, ε, το αναλάβατε. Από το Connecting Europe Facility έχουμε χάσει χρήματα και από τον ορίζοντα για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έγινε μια πρόταση για την ευρυζωνικότητα και μόνο να δοθούν περισσότερα χρήματα. Τώρα γίνονται οι επόμενες συζητήσεις με τον κύριο Κατάινεν για επέκταση του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν έχει έρθει η ώρα να ε, επικεντρωθούμε κάπου. Η Ευρώπη δεν μπορεί να ασχολείται με τα πάντα. Θα πούμε, θα αφιερωθεί στην ψηφιοποίηση και στην ευρυζωνικότητα. Γιατί ε, τώρα ε, προσπαθούμε πάλι να ρυθμίσουμε τα πάντα. Αν έχουμε χρήματα από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ε, μάλλον από τον ορίζοντα 2020, δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε στην ευρυζωνικότητα. Γιατί Μάλλον φεύγουν χρήματα από το τομέα αυτό αυτή τη στιγμή παρά μπαίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. σε αυτό το τομέα ειδικά είναι σαφίστατη η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής δράσης. Εδώ λοιπόν μπορούμε πραγματικά να διασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του τομέα. Ιδιαίτερως θα ήθελα να θίξω ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις ε, ψηφιακές εγκαταστάσεις και την, ε, την επίκουσα ανάγκη διασύνδεσή του είναι κάτι το οποίο ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι και αναφέρεται γενικά από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Είναι θεμελιώδη σημασία. Δεύτερο στοιχείο για ε, τον κλάδο. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε προποθέσει, ιδίω ό,τι αφορά την ε, κυβερνοασφάλεια, αλλά όχι αποκλειστικά και μοναδική, σε ό,τι αφορά τι ε, νέε βιομηχανίε και νέε κατασκευαστικέ ε, τεχνολογίε και πώ αυτέ θα συνδεθούν με την αλυσίδα εφοδιασμού. Και εκεί αυτά συνδέονται και με στήματα ασφάλεια. Και τέλο, σε ό,τι αφορά τι δεξιότητε και τι θέσει απασχόληση, που είναι κρίσιμη σημασία και για του πολίτε μα πρέπει να στοχεύσουμε σε δύο τομείς. Διαβίου μάθηση, αλλά και το φιλετικό το μάλλον το χάσμα μεταξύ των δύο φίλων. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα διάσταση του φίλου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε και για την δέσμη μέτρων. Για το DSM για ε, την ψηφιακή νέα αγορά είχαμε παραπονεθεί ότι θέλαμε να συμμετάσχει και ο κλάδος και είναι πολύ καλό που συμβαίνει αυτό τώρα. Πολύ θετική σημερινή συζήτηση, το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, πώς θα ψηφιοποιηθεί η Ευρώπη. Υπάρχουν ορισμένες καινοτομίε που θεωρώ ότι θα πρέπει να θέσουμε και να εξετάσουμε διαφορετικά. Και εγώ, επειδή είμαι από τη Φιλανδία, ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένε καινοτομίε που θα πρέπει να μα απασχολούν ιδιαίτερω, όπω ε, αυτέ που αφορούν την ε, τιμολόγηση. Τώρα στην Ευρώπη χρησιμοποιώ τα κινητά δεδομένα, αλλά τα πληρώνω όλα. Όμως στη Φιλανδία υπάρχουν συγκεκριμένα πακέτα ε, απεριόριστης χρήσης ε, όταν κάποιος επιλέξει μία ταχύτητα. Άλλοι, ας πούμε, θέλουν να πάρουν ένα φτηνό ε, πακέτο με χαμηλή ταχύτητα. Εγώ όμως, επειδή χρειάζομαι μεγάλο όγκο, ε, χρειάζομαι υψηλή ταχύτητα και μου κοστίζει 30-40 ευρώ το μήνα και μπορώ να σου πλήσω όσα δεδομένα θέλω στο κινητό μου. Και ε, πήγα από τη Λαπωνία στο Ελσίνκι, χίλια χιλιόμετρα και ήμουνα συνεχώς συνδεδεμένη. Δεν υπήρξε ποτέ διακοπή. Και πολλέ επιχειρήσει λένε ότι αυτό είναι ε, κερδοφόρο. Επομένω, μπορούμε να εξετάσουμε και τέτοιε λύσει ε, απρόσμενε. Πρόεδρο, δεν ξέρω αν θέλει κάποιο άλλο να πάρει τον λόγο, γιατί έχουμε φτάσει στο τέλο του καταλόγου μελητών. Παρακαλώ, ο κύριο Κέλλη. Ναι, εν συντομία. Στι μεταφορέ. ιδίω ό,τι αφορά κατηγορίες λεωφορείων και το καθεξής, ε, φορτηγών. Ξέρω ότι το κόστος είναι τεράστιο, η εξοικονόμηση χρόνου ε, θα ήταν πολύ σημαντική, αλλά και η εξοικονόμηση σε εκπομπές δεξιδίου του άνθρακα και ο χρόνος οδήγησης και μεταφοράς. Δεν ξέρω, μπορούμε να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε πάρτε μια βαθιά ανάσα και έχετε να απαντήσετε 57 ερωτήσεις. Μάλλον αδύνατον, αλλά προσπαθήστε. Ε, με το ITU είμαστε σε στενή επαφή, συμμετέχουμε και σε διασκέψεις συχνά. Μόλις το roaming η περιαγωγή στην Ευρώπη γίνει νόμος, θα περάσουμε και στο επόμενο βήμα θα κάνουμε την νομοθετική πρόταση που ήδη έχουμε εξαγγείλει. Είναι η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών αυτή στη Γενέβη. Ε, το χρόνο το Μάιο καλό θα ήταν να ε, έρθουν όλα αυτά στην αγορά για να εφαρμοστούν. Και εφόσον και αυτή τη στιγμή έχουμε ευρωπαϊκή περιαγωγή, θα το θέσουμε και ως θέμα στις εταιρικέ σχέσεις και συνεργασία που έχουμε με άλλες περιφέρειες του κόσμου και για τη γενική τυποποίηση. Από το χρόνο το Μάιο δηλαδή, ε, ελπίζω να ε, είμαστε επιχειρησιακοί. Δεύτερον, για το 5G θα βάλουμε εμείς δικά μας πρότυπα, αλλά έχουμε μια κοινή δήλωση με την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, ήδη υφίσταται και ε, διαπραγματεύομαι τώρα και με άλλους με τις Ηνωμένε Πολιτείε για να έχουμε ένα ιστό αράχνης ας πούμε με τα σημαντικότερα άλλα παγκόσμια δίκτυα ε, ε, για να μπορέσουμε στα πλαίσια της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών να εργαστούμε πιο εύκολα και ε, στην αρχή της επόμενης δεκαετίας το 5G να έχει παγκόσμια πρότυπα για να μπορούν αυτές οι υπηρεσίες και οι μεταφορές δεδομένων να γίνονται ψηφιακά και τυποποιημένα. Τώρα, ρωτήσατε για σημαντικά έργα που σας ενδιαφέρουν. 30 με 40 δις το χρόνο θα μπορούσαμε να χρειαστούμε και αυτός είναι ο συνολικός γεωργικός προϋπολογισμός για αυτά τα έργα και μόνο. Δεν τα έχουμε όμως. Έχουμε μονοψήφιο αριθμό δισεκατομμύρια για τα ψηφιακά. Αν τα προσθέσω όλα, θα θρήσω. Ευχαριστώ τον κύριο Έλερ που μίλησε για τον ορίζοντα 2020. Γίνονται κάποια πράγματα συμπληρωματικά, αλλά είπατε για το Connecting Europe η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 9,6 δις και έγινε 1 δις. Τώρα, 1 δις τι να το κάνω, δεν χρειάζεται καν να μπω ε, στη ε, ε, συζήτηση να αρχίσω κανένα εγχείρημα γιατί δεν με φτάνει αυτό ούτε για τη βενζίνη μου. Για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το σχέδιο Juncker. Αυτό λειτουργεί πρώτα απ' όλα με κάλυψη κινδύνου και λιγότερο με μετρητά. Ανάληψη κινδύνου. Υπάρχει ένας, ένα χωριό στην Ήπεθρο με τρεις οικισμούς. Ε, η οπτική είναι, δεν είναι ε, ρίσκο, είναι απώλεια δεδομένη. Ξέρουμε ότι έχουμε 30 συμβαλόμενα μέρη και μια επένδυση, ε, προκήρυξη διαγωνισμού και περίπου 40% ε, ε, αυτό που χρειάζεται είναι μετρητά. Αυτό δεν το έχει το έφηση και ο κίνδυνος είναι 100%. Είναι εγγυημένη απώλεια, δεν είναι ρίσκο. Γι' αυτό δεν, δεν καλύπτεται αυτό από το ΕΦΣΙ. Με πακέτο θα μπορούσε να καλυφθεί, αλλά στην ευρυζωνικότητα, εκεί που δεν είναι κερδοφόρο αυτό το εγχείρημα, αυτό που βοηθάει μόνο είναι ε, η χρηματοδότηση από ε, δημόσια κονδύλια, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά, είτε είναι περιφερειακά, εθνικά, τοπικά, από κάποιο κρατικό κουρβανά. Ε, όταν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι πολύ σημαντική ε, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εμπειρία στην αξιολόγηση και στην έγκριση τέτοιων προγραμμάτων. Τώρα, για την οικονομική ενίσχυση Ποια είναι τα πιο σημαντικά για μας. Αυτή η ψηφιακή κόμβη, τα hubs, είναι τριψήφιος αριθμός εκατομμυρίων εδώ. Θέλουμε σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης να υπάρχουν κέντρα συμβουλευτικά. Είτε αυτά είναι δημόσια, είτε είναι σε ένα κάποιο επιμελητήριο ή σε έναν άλλο φορέα. Διότι πιστεύουμε ότι μικροί ε, τεχνίτες, επαγγελματίες, ε, ένας αρτοπιός που έχει τρεις φούρνους, ξέρω εγώ, θα πρέπει πρώτα απ' όλα για θέματα ψηφιακά να έχουν ε, ε, παροχή συμβουλών. Υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και τις μικρομεσαίες. Αυτό πρέπει να καλυφθεί. Χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια για τη συγχρηματοδότηση υπερυπελογιστών για να μπορέσουμε να έχουμε ε, υψηλής απόδοσης ε, υπολογιστές στην Ευρώπη για όλους τους Ευρωπαίους. Για το ερευνητικό νέφος επίσης θα χρειαστούν πολλά χρήματα, το cloud εκεί. Και επίσης θέλουμε να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό νέφος ε, έτσι ώστε να έχουμε συνεργασία με, ένα διάφορα Ινστιτούτα κοντά στην οικονομία, όπως είναι στη Γερμανία το Ινστιτούτο Fraunhofer, και όλα τα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και για τη βιομηχανία και τις εταιρείες που κάνουν έρευνα. Να υπάρχει μια βάση δεδομένων, προσβάσιμη για όλους, ε, δημόσια, ανοιχτή, δωρεάν και να μπορεί να υποστηρίζει ε, ψηφιακά την έρευνα. Έρχομαι τώρα στα προσόντα, στις δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτιση, μετεκπαίδευση. Γιατί έχουμε αυτό το ψηφιακό χάσμα. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν βασικές γνώσεις ψηφιακές, κοινωνικά μέσα δικτύωση, social media, έχουν διάφορες εφαρμογές που τις χρησιμοποιούν ενεργά, από συσκευή σε συσκευή, ε, κάνουν ψηφιακή παραγωγή και κάποιοι που δεν έχουν αυτές τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Αυτό είναι το ψηφιακό χάσμα. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, η κατάρτιση, η μετακπαίδευση δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα αρμοδιοτήτων. Και αυτές τις μέρες που κυκλοφορούν διάφορα δημοψηφίσματα και ε, δεν θέλει να αναγνωρίσει κανένας τίποτα σε εμά τους ευρωκράτες, είμαι κάπως επιφυλακτικός. Αλλά εργαζόμαστε εκεί. Ε, ε, καλέσαμε τους υπουργούς έρευνας και επιστήμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο έχουμε 160.000 που χρειαζόμαστε στην πληροφορική. Φυσικούς, πληροφορικάριους ε, ε, και διαφόρους ε, που ειδικεύονται στην πληροφορική. Δεν αρκούν οι θέσεις που προσφέρονται στα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή για φοιτητές και θα πρέπει να συμφωνήσουμε ε, με τα πανεπιστήμια και τους αρμόδιους φορείς που καμιά φορά ε, είναι υπουργοί ε, αρμόδιοι παιδείας και επιστήμης και εθνική και περιφερειακή έτσι ώστε να αυξηθούν οι θέσεις στα πανεπιστήμια και την επόμενη δεκαετία να καλυφθούν οι ανάγκες που θα δημιουργηθούν στην αγορά εργασίας. Και για τις δεξιότητες και τα προσόντα έχουμε την πρόθεση να έχουν μια ευρεία συμμαχία ε, και εκεί να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες, τα συνδικάτα, ε, τα ευρωπαϊκά, οπωσδήποτε. Είναι κοινή προσπάθεια, είναι κοινό εγχείρημα και κοινό μέλημα των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων και των δικών τους συνδικαλιστικών εκπροσώπων και οργανώσεων. Το cloud computing, το υπολογιστικό νέφος, νομίζουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να καταστεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Προσοχή όμως. Δεν θα πρέπει να αποκοπεί η Ευρώπη. Είναι παγκόσμιο αυτό το εγχείρημα. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια που κάνουν οι ΗΠΑ ή η Κορέα που προσφέρουν ε, δυνατότητες αποθήκευσης ή επεξεργασίας δεδομένων και για ευρωπαϊκά ε, δεδομένα και εταιρείε και επιχειρήσεις. Η προστασία όμως των δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων πρέπει να είναι ακριβώς δεδομένη με συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές. Και αντίστροφα, όταν ε, υπάρχει μια υπηρεσία cloud στην Ευρώπη, είτε είναι ευρωπαϊκή εταιρεία, είτε είναι ξέρω εγώ, μια κοινοπραξία της Microsoft με το systems η Microsoft επενδύει στην Ευρώπη σε υπηρεσίες cloud έτσι ώστε με την εμπιστοσύνη ότι θα εφαρμοστεί και πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων. Δημιουργεί νέφη που δεν θα δημιουργούσε στην Αμερική ή που δεν θα υπήρχε τόση προστασία. Έχουμε λοιπόν cloud της Microsoft στην Ευρώπη ε, που υπόκειται μόνο στο ευρωπαϊκό δίκτυο ή μήπω οι μυστικέ υπηρεσίε των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν και εδώ πρόσβαση. Όχι, αυτό το αποκρούουμε ε, στεναρά, διότι στην ευρωπαϊκή επικράτεια ισχύει ε, ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων και όχι να αλωνίζουν μυστικέ υπηρεσίε άλλων χωρών. Θα κάνουμε και θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε μαζί σας, έτσι, ώστε να επιταχύνουμε τις διαβουλεύσεις για τα ψηφιακά. Κυρίες και κύριοι, στη Γεωργία, όταν συζητάτε για τη 17η πλευρά, ξέρω εγώ, ε, ε, στο χείριο κρέας ε, και πώς εκτρέφονται οι χείροι, έχετε χρόνο, μπορείτε να το συζητάτε 10 χρόνια. Όταν συζητάμε όμως για τη φορητότητα των αριθμών, για τα ψηφιακά και χρειαζόμαστε πέντε χρόνια από την πράσινη βίβλο μέχρι να γίνει λευκή βίβλος, συζητήσεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις υπηρεσίες, απόφαση, κοινοβούλιο, συμβούλιο, τριμερής διάλογος και εφαρμογή σε εθνικό δίκαιο, πέντε χρόνια αργότερα η τεχνολογία και οι συμμετέχοντες έχουν πάει μια γενιά πιο κάτω. Και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα έχει κανένα κύρος έτσι. Θα πρέπει να είμαστε κοντά στις εξελίξεις και να αποφασίζουμε πολύ γρήγορα. Διαβούλευση σε βάθος βέβαια, αλλά ταχεία. Και ε, οι τηλεπικοινωνίε είναι ένα παράδειγμα εδώ και είμαι σε στενή επαφή με τι δύο επόμενε προεδρίε του Συμβουλίου, που είναι η Σλοβακία και η Μάλτα. Μέσα σε ένα χρόνο η πρόταση ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να εφαρμοστεί και να ισχύει ω δίκαιο. Ρωτήσατε τι έγινε στην Αυστρία, στο ΛΕΧ, στο φόρουμ. Κάποτε υπήρχε ένας καγκελάριος, που ε, ο Σούσελ στην Αυστρία, που δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ στο ΛΕΧ της Αυστρίας. Αυτό στη συνέχεια ε, ε, έγινε, κάπως αδράνησε, ε, γίνεται στο Φόραλμπερκ της Αυστρίας, το ΛΕΧ, εγώ, είναι από τη δική μου αιγίδα, μπορούμε να σας στείλουμε τα απορίσματα των τεσσάρων πάνελ ε, τις επόμενες εβδομάδες και από τους συνεργάτες μου και από μένα μπορείτε να μάθετε ό,τι θέλετε για το πώς πήγε εκεί το φόρουμ, τι συζητήσαμε, πώς το προετοιμάσαμε και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το 2017 το επόμενο. Μπορώ να σας απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Κατά τα άλλα, υπάρχει ε, το Digital Agenda Assembly, μια συνέλευση που θα γίνει φέτος στην Πρατισλάβα. Είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερομένους, βουλευτές, πολίτες, όποιος θέλει μπορεί εκεί να έρθει να γίνει η συνέλευση αυτή, η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο κύριος Άνσιπ και εγώ ετησίως συμμετέχουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Μια τελευταία ερώτηση. Το vectoring είναι ένα γερμανικό ζήτημα. Αλλά είναι ενδεχομένως και ένα προσχέδιο ε, για μελλοντικές ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και από τις 7 Απριλίου που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα είναι και θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η γερμανική Deutsche Telekom έχει ζητήσει για τα τελευταία 500-600 μέτρα να αυξηθεί η ε, χωρητικότητα με το vectoring. Αυτό υπάρχει ως δυνατότητα. Η αρμόδια αρχή έκανε πρόταση Είναι 63 σελίδες και τώρα θα πρέπει να το ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι αυτό το vectoring, η ανισματική διακοπή. Εγώ ε, θα πρέπει να κάνω τι, να έχω ένα διαιτητικό ρόλο, είμαι και εδώ επιφυλακτικό. Μέχρι τις 10 Μαΐου πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις μας και τρεις είναι οι στόχοι. Το vectoring αυτό κατά αυτό είναι μια τεχνολογία έτσι ώστε βράχει πρόθεσμα να αυξηθεί η δυνατότητα χωρητικότητας υφισταμένων δικτύων. Αλλά δεύτερον, δεν θέλουμε έτσι να επανέλθουμε σε ένα μονοπόλιο ξανά και επίσης δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο οι ε, επενδύσεις ε, που έχουν ξεκινήσει για τις οπτικές ίνες να ε, καταστούν ασύμφορες. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε αυτά που μας απασχολούν, ε, αν έχουν απαντηθεί όλα με τις συγκεκριμένες τεχνολογίες, αν πρέπει να περάσουμε σε δεύτερη φάση του άρθρο 7 ή 7α της οδηγίας για τις τηλεπικοινωνίες, χρειάζονται δύο ή τρεις μήνες για την εφαρμογή τους. Έχω λάβει επιστολή από διάφορους βουλευτές, την κυρία Κάμερβερτ και άλλους, Είμαι στη διάθεσή σας για συνομιλίες ε, το επόμενο διάστημα, τις επόμενες τρεις εβδομάδες ή δύο-τρεις μήνες ε, για να κάνουμε συζητήσεις κατηδία. Και πραγματικά πιστέψτε με, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα, γιατί έχουμε και μεγάλους ανταγωνιστές και μικρότερους τοπικούς και γίνονται και πολλές ερωτήσεις και ε, στη Γερμανική Βουλή, την Bundestag. Τελειώνω. Η συμφωνία συνασπισμού που έχει η γερμανική κυβέρνηση ως βάση ε, ε, συζήτησης και, και λειτουργίας κυβέρνησης κάνει το θέμα ακόμα πιο ευαίσθητο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Ήταν αδύνατο να βρούμε μια μισή ώρα αυτή τη φορά για τη συνάντησή μας με τον ε, Επίτροπο Έτιγκερ. Σίγουρα η μία ώρα δεν φτάνει. Την επόμενη φορά όμως ε, θα έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Μια μέρα, ναι, καλύτερα θα ήταν, έχετε δίκιο. Να έχουμε μια ολόκληρη μέρα στη διάθεσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που απευθύνατε σε όλους μας για τη συνδιάσκεψη στις 25 Απριλίου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, για την ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Εσείς θα ηγηθείτε, η κυρία Μπενικόφσκα και ο κύριος Μόιδας, τρεις επίτροποι λοιπόν από κοινού, υπό την Ολλανδική Προεδρία, στο ανώβερο από ό,τι κατάλαβα. Και θα παρίσταται και υπουργοί σε ύψιστο λοιπόν επίπεδο η συνδιάσκεψη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστούμε που ήσασταν και εδώ μας σήμερα μαζί μας. Um, Συνάδελφοι, ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Επόμενο σημείο στην εμείς διάταξη Φαντάζομαι έχετε όλοι τις κάρτες σας μαζί σας. Και τώρα θα κάνουμε έναν δοκιμαστικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Απαντήστε αν είστε έτοιμοι. Υποθέτω είστε όλοι έτοιμοι. Πέρας. Εντάξει. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, συνάδελφοι, μία νέα συμφωνία για τους ε, καταναλωτές ενέργειας. Η συγκήτρια κυρία Γκρίφιν. Θα αρχίσουμε αμέσως. Στη 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Τμήμα 1 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 18. Τμήμα 1. Ένας παραπάνω στους σοσιαλιστές. Δύο παραπάνω. Πέρας. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα καταπίπτει. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Η 19. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται από ό,τι βλέπω. Εντάξει. Τροπολογία 26 με προφορικές τροπολογίες. Δεν ξέρω αν ε, διαφωνεί κάποιο ή θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Τροπολογία 26 με τι ε, προφορικέ τροπολογίε λοιπόν. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 35. Υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Για την 35. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημαντική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές. Να την ελέγξουμε. Τη 43. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, μάλλον τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε την τροπολογία 65 Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 82 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 82 πέρας εγκρίνεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε πέρας εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, ναι, να ελέγξουμε. Εντάξει, βεβαίω. Την 102 λοιπόν ελέγχουμε. Πέρα. Εγκρίνεται. Να ελέγχουμε λοιπόν πιο συχνά. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 103. Πέρας. Εγκρίνεται. 26, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τη 226. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι συνάδελφοι εδώ στα αριστερά, παρακαλώ να ψηφίζετε. Εγώ έκανα λάθος, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Να σας βλέπω, παρακαλώ. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εκρίνεται. Βλέπετε τώρα. 195. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Την 195. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τη 13α. Πέρασε. Εγκρίνεται. 128. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 153 μήμα 2 υπέρ Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Την 153 τμήμα 2. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ με την προφορική τροπολογία βέβαια. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να πάρει τον λόγο. Εντάξει. 201. Χωρίς την τροπολογία. Γιατί μία πολιτική ομάδα αρνείται την τροπολογία. 201 τροπολογία χωρίς την προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. 201 χωρίς την προφορική τροπολογία λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται. Η θεμαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 223 τμήμα 2 υπέρ, κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 7 τμήμα 2 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2.45 κατά αποχές σας ελέγξουμε τη 2.45 ελέγχουμε πέρας εγκρίνεται. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 2.52. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.53 υπέρ. κατά, αποχές. Μάλλον το ίδιο θα είναι, οπότε εγκρίνεται. 2.54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.56 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε τη 2.56. Πέρασε. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. 2.57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Πέρασε τη 2.57. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 303, 13 μάλλον, υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε την 313. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.15 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά 3.15. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 356 υπέρ κατά ελέγχουμε την 356 πέρας Εγκρίνεται. Συμβαστική 35 Περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 371 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 380 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε. 380. Πέρας. Απορρίπτεται. 381 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε και πάλι την 381. Πέρας. Απορρίπτεται. 388 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε και την 388. Απορρίπτεται. 428 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 381 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.90 υπέρ κατά να την ελέγξουμε την 3.90 πέρας απορρίπτεται 3.91 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε και πάλι την 3.91 Έγκρινεται αυτή τη φορά. 34. Υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 34. Πέρας. Εγκρίνεται. 37 συμβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έχουμε 5 τροπολογίες από την 4.19 έως την 4.23 που είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε από κοινού λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά ας την ελέγξουμε. Ελέγχουμε. Πέντε τροπολογίες από κοινού. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνονται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ένα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο σύνολο της έκθεσης για τη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας, πέρας, εγκρίνεται συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και σε όλους τους κοιόδης και όλους εσάς για τη σκληρή δουλειά που έγινε σε αυτήν την Επιτροπή. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο, συνάδελφοι. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Σημείο 13. Ανταλλαγές απόψεων με τον ΕΝΙΣΑ. Ο τομέας ασφάλεια στην κυβερνοχώρο στο πλαίσιο μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη ψηφιακή βιομηχανική πρωτοκαθεδρία. our uh, dear colleagues, Teresa Ma Petra, well, please. Συνάδελφοι, Τερέζα, Πέτρα, παρακαλώ μην κάνετε πηγαδάκια. Colleague coordinator, done. okay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 Uh, on Εξ ονόματος όλων συγχαίρω και πάλι την Τερέσα Γκρίφιν. Μπορούμε έτσι να κλείσουμε τους εορτασμούς. Συγχαρητήρια, αλλά να τελειώνουμε σιγά σιγά. Συναδελφοί, ας ε, στραφούμε τώρα στο θέμα μας. Ανταλλαγή απόψεων με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Η ασφάλεια στην κυβερνοχώρο ως ε, μια οικονομική ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ούντο Χέλμπρεχτ είναι μαζί μας, ε, διευθυντής του ΕΝΙΣΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού λοιπόν, για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Εξαιρετικά σημαντικό ο οργανισμός αυτός. Υπενθυμίζω ότι στις 19 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ε, ψηφιακή βιομηχανική πρωτοκαθεδρία. Μια ειδική δέσμη μέτρων λοιπόν για την Επιτροπή μας. Γιατί εμάς μας απασχολούν τέτοια ζητήματα ε, ψηφιακής βιομηχανικής πρωτοκαθεδρίας στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να σας πενθυμίσω ότι το θέμα της ασφάλειας στην κυβερνοχώρο είναι θέμα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για τα μέλη της Επιτροπής μας. Είναι και στον τομέα των αρμοδιοτήτων μας. Όμως, μέχρι τώρα σημείο εστίαση ήταν περισσότερο η διασφάλιση της ασφάλειας στην κυβερνοχώρο. Σήμερα θα αλλάξουμε σημείο εστίαση και θα στραφούμε προς ε, τις οικονομικές δυνατότητε που μας ε, παρέχει ο τομέας της ε, ασφάλειας στην κυβερνοχώρο. Γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε και νέους κλάδους της βιομηχανίας βάσει Τη πάλης μας αυτή ε, και των προσπαθειών που καταβάλουμε για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Κύριε Χιάνμπρεχτ, έχετε το λόγο για τα εισαγωγικά σα σχόλια. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σα. Σα Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι χαρά και τιμή μου που είμαι σήμερα εδώ. Θα σας μιλήσω για το τι κάνουμε στην, στον οργανισμό ΕΝΙΖΑ, καθώς και για την κοινή ψηφιακή αγορά ως μέσο για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και οικοδόμησης ε, και για την οικοδόμηση ε, εμπιστοσύνης. Εάν είχαμε την ομιλία του Επιτρόπου Έτιγκερ ήδη και ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε, γι' αυτό και είναι καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για την ασφάλεια. Θα σα μιλήσω για τρία θέματα. Καταρχά τι εννοούμε σήμερα όταν λέμε τη λέξη digital, ψηφιακό, τι είναι σημαντικό για την βιομηχανία και ε, επίσης ε, τι εννοούμε όταν λέμε πρωτοκαθεδρία της Ευρώπης. Αν δούμε Καταρχάς, ε, ο ψηφιακός κόσμος αγκαλιάζει κάθε κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Έχουμε ηλεκτρονική τραπεζική, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική παιδεία ή ηλεκτρονικά από όλα και θέλουμε όλα αυτά να λειτουργούν σε έναν ανοιχτό ασφαλή ε, κύβερνο χώρο. Βλέπουμε την εφή κατα, κα, κατασκευή, το ίντερνετ των πραγμάτων καθώς και κρίσιμες υποδομές για του, το, τους υπολογιστές. Η πρόκληση, αν δει κανείς αυτό τον ψηφιακό κόσμο, ε, είναι ότι έχουμε αλλαγές στα επιχειρηματικά μοντέλα, πράγμα που σημαίνει με τη σειρά του ότι έχουμε διακοπτό και διαφορετικά ε, μοντέλα. Ε, δηλαδή αν έχουμε τις παραδοσιακές ε, αλυσίδες αξία όπου παράγει κανεί ένα προϊόν δηλαδή και το πουλάει, τώρα έχουμε ένα σωρό πλατφόρμες όπου πάνω από αυτή την κατασκευή δημιουργούνται επιχειρηματικά μοντέλα. Ας πούμε αν δούμε την Uber δεν χρειάζονται πια τα ταξί. Αν μιλάμε για τα ευφύ τηλέφωνα, Χρειάζεται ένα αυτοκίνητο με τέσσερις τροχούς, το οποίο ελέγχεται μέσω του τηλεφώνου. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε στον ψηφιακό κόσμο στην Ευρώπη, έτσι ώστε τα έσοδα αλλά και οι θέσεις απασχόλησης να μένουν εδώ. Πρέπει λοιπόν να αγκαλιάσουμε αυτή την πρόκληση να τη συζητήσουμε. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι πώς θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη σε όλα αυτά με το πολιτιστικό μας υπόβαθρο εδώ στην Ευρώπη, πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα εμπιστευόμενοι τα στοιχεία και τις διαδικασίες. Και αν το εξετάσουμε αυτό, τότε έχουμε επίσης και στην ιδιωτική μας ζωή ε, να μας απασχολήσει το θέμα. Μιλάμε για ευφύη τηλέφωνα, ευφύης πόλης, ε, όπου υπάρχει σύγκληση διαφόρων τομέων, όπως ε, ε, τον αυτοματοποιημένο δημόσιο τομέα, στις μεταφορές, στις παρακολούθηση. Ένα σωρό πράγματα. η νέα γενιά τα χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντοτε υπογραμμίζει την ε, ψηφιακή μεταμόρφωση. Μιλάμε λοιπόν εδώ για τα, πολύ για δεδομένα. Αν δούμε τα δεδομένα από την άποψη της ε, διάρκειας ζωής των δεδομένων, τα δεδομένα παράγονται, ε, υπόκειται σε επεξεργασία, κάποιες φορές παραμένουν για πάντα. Και πώς αυτά συνδέονται με τα επιχειρηματικά μοντέλα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη και τα δεδομένα, θα πρέπει να δείτε ένα έγγραφο θέσεων που δημοσιεύσαμε πριν από κάποιες ομάδες όσον αφορά την κρυπτογράφηση ας πούμε, είναι σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη σε τον οικονομικό κόσμο και να έχουμε ασφαλή επιχειρηματικά μοντέλα και διαδικασίες επεξεργασίας ε, δεδομένων. Ας πούμε, αν θέλει κανείς να πάει στην ηλεκτρονική υγεία, αν θέλει να έχουμε ε, τα αρχεία και τους φακέλου των ασθενών δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε μόνο αν υπάρχει μια ε, μεγάλη εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Τώρα τα big data είναι τεράστιο αριθμός και όγκο στοιχείων που γεννώνται σε ολόκληρο τον κόσμο και αν κανείς πάει σε ένα επιγραμμικό μαγαζί θα δει ε, το μήνυμα του που λέει και άλλοι αγόρασαν το ίδιο για να σας επηρεάσει και να ε, το αγοράστηκε. και και δείτε τα διάφορα στατιστικά μοντέλα είναι κάτι πολύ εύκολο. Ε, από πραγματικές πληροφορίες δηλαδή οι εταιρείες, οι πολίτες, οι χρήστες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και να ε, κατευθυνθούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς γίνονται όλα αυτά. Τώρα ε, cloud computing. Ε, εμείς στην ΕΝΙΖΑ το έχουμε αυτό εξετάσει, έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε την ασφάλεια στην ε, τεχνολογία. Δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά σήμερα βρίσκουμε διαδικτυακούς χώρους όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμός εταιριών που αποκαλύπτει στοιχεία, αποκαλύπτει πώς λειτουργεί με αυτά. Η πρόκληση είναι να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση ώστε ο κόσμος να γνωρίζει τέτοιες, πού υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Ε, επίσης θέλω να αναφέρω για αυτό το πρώτο τμήμα του κανονισμού προστασία ε, τη ψηφιακή αγορά θέλω να πω ότι είναι ευπρόσδεκτο, αλλά θέλω επίση να παρατηρήσω ότι αν θέλουμε αυτό να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι τεχνολογίε, να αναζητήσουμε τι τεχνολογίε που εξασφαλίζουν και ασφαλίζουν την εφαρμογή. Όταν λέμε λοιπόν για ιδιωτικότητα και σχεδιασμό, ε, σημαίνει τη χρήση πολλών τεχνολογιών ε, Χιλιάδες νέος κόσμος χρειάζεται για αυτή την αρχές ε, προστασίας των δεδομένων. Το θέμα είναι αν, υπάρχει, ε, αν υπάρχουν οι δεξιότητες ε, για την τεχνολογία αυτή και κατά πόσο υπάρχουν τα απαραίτητα στελέχη τόσο στην κυβερνητικό μηχανισμό όσο και στις επιχειρήσεις για να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης η βιομηχανία. Έχουμε πρωτοβουλίες όπως ε, η καινοτομία για την μεταπίση για τις μικρομεσαίες, το Age 2020, τον ορίζοντα 2020, το διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και τα λοιπά διάφορα μέσα και έρευνα και, ε, ε, έρευνα και ανάπτυξη νέας γενιάς. Θα πρέπει να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία, τι κάνουμε μάλλον με τα στοιχεία των ασθενών, του φακέλου των ασθενών. Θέλουμε να υπάρχει ένα τομέα ηλεκτρονικός για την υγεία που θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία, θα ωφεληθεί ο ασθενής, τα, τα νοσοκομεία για τις ε, επεμβάσεις, αλλά υπάρχουν ζητήματα γιατί δεν υπάρχει ελεύθερη ροή των στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που είναι ξεπερασμένοι, δεν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες ε, του cloud, του νέφους. Είναι μια τεράστια αγορά στην Ευρώπη γιατί η υγεία Μάλλον υπάρχει αντίσταση γιατί η υγεία είναι τοπικό, τοπική ε, υπόθεση. Θέλω να αναφέρω δύο σημαντικούς στόχους στρατηγικής φύσης που συζητάμε στο Διοικητικό μας Συμβούλιο. Είναι η οικοδόμηση κοινοτήτων και δυνατοτήτων. Το κάνουμε αυτό σε συνεργασία με την Κομισιόν, σε ένα project ε, ιδιωτικού με ε, ε, δημόσιο τομέα συμπεριλαμβάνονται και οι μικρομεσαίες, διοργανώνουμε διάφορα εκδηλώσεις και έτσι ε, οικοδομούμε ε, δυνατότητες σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε άλλους τομείς με τη στήριξη, στηρίζουμε μάλλον τα κράτη-μέλη. Τώρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την πρωτοκαθεδρία, κάνουμε αυτά δύο χρόνια, κάνουμε ευρωπαϊκές ασκήσεις, θα το κάνουμε και φέτος το φθινόπωρο, όπου θα συγκεντρώσουμε εκατοντάδες διαφορετικούς θεσμούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς, ώστε να αναζητήσουμε σενάρια και την στεναρότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών υποδομών. Θα ήθελα επίσης να τονίσω αυτό που ήδη ανέφερα, Ότι δηλαδή αν δούμε αυτό το τομέα δεν υπάρχει λογοδοσία, δεν υπάρχει ευθύνη όπως υπάρχει σε άλλους τομείς. Ναι, ορισμένες ε, βιομηχανίες δεν τους αρέσει το, η, η, λογοδοσία, η ευθύνη μάλλον για το λογισμικό. Το θέμα όμως είναι και πώς και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Αν μιλάμε για τη διασύνδεση των αυτοκινήτων, ας πούμε, μπορεί να είναι αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά σε άλλους τομείς είναι δύσκολο να βρούμε τη ρίζα του προβλήματος και να μπορέσουμε να καλύψουμε και να πιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που αναπτύσσουν ε, καθαρά μόνο λογισμικό. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι τώρα έχουμε κλείσει τα 12. Εξετάζουμε διάφορα μοντέλα και το μέλλον αυτών, καθώς και τις ευκαιρίες. Γι' αυτό και δημοσιεύουμε πολλά έγγραφα. Είμαστε δεσμευμένοι στην συνεργασία. Καλωσορίζουμε τις, ε, τις ε, πρωτοβουλίες της Επιτροπής και θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, κύριε Βουζέκ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρέμβω και να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κύριε Καφεντά, μπορούμε τώρα να περάσουμε στους προσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μπόνι εκ μέρου ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Α, συγγνώμη, κύριο Έλερ. Δεν το ήξερα. Ο κύριο Έλερ. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Η Επιτροπή εξετάζει τον προπολογισμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μιλητή, γιατί νομίζω ότι χωρί τη δική του ε, συμβολή ενδεχομένω ε, να μην υπήρχε πλέον ο σε αυτό ο οργανισμό και ούτε όλη αυτή η συζήτηση στην οποία έχει συνεισφέρει. Νομίζω ότι πραγματικά έχει επιδείξει μεγάλη αφοσίωση και θα ήθελα να του πω ότι εκτιμούμε αυτή του την προσφορά. Έχει κάνει πολλά για να στηρίξει τον ΕΝΙΣΑ και νομίζω ότι μπορούμε να ασφάλεια να πούμε ότι χωρί εσά δεν θα είχαμε όλε αυτέ τι εξελίξει. Δύο ερωτήσει τώρα. Πρώτον, γίνεται το λένε και πιο σαφέ ότι η πρώτη γραμμή υπεράσπιση κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι η δημόσια δράση. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα αντικατοπτρίζεται και θα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις, ε, στη βιομηχανία δηλαδή και ο ΕΝΙΣΑ έχει έναν πολύ σαφώ καθορισμένο ρόλο, γιατί τα κράτη-μέλη ήθελαν να περιορίσουν ε, τις αρμοδιότητες του ΕΝΙΣΑ, ιδίω ό,τι φορά τη δημόσια σφαίρα. Υπάρχει πολύ σαφώ ορισμό του ρόλου του ΕΝΙΣΑ και του συντονισμού ε, των προσπαθειών που καταβάλλονται στον κλάδο. Όμω, πώς έχει η κατάσταση σήμερα, μετά από μια δεκαετία, τι πρόοδο έχουμε σημειώσει ως προς την τυποποίηση. Μιλούμε πλέον για ελάχιστα πρότυπα, απόλυτα πρότυπα. Πόσο ασφαλείς είναι οι νέες υπηρεσίες και σε ποιο βαθμό έχουν ενσωματώσει ε, την ε, ασφάλεια εκ του σχεδιασμού οι νέες υπηρεσίες. Υπάρχει επίσης και το ζήτημα της ε, δέσμευσης και εμπλοκής ε, του κλάδου μας ε, στην κυβερνοασφάλεια. Και μετά σε ό,τι φορά την παράταση της εντολής σας, ξέρω ότι τώρα οι λειτουργίες σας εδράζονται στην Αθήνα, αλλά βλέπω ότι το πρόβλημα γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Επομένω, τι χρειάζεται ο ΕΝΗΣΑ και από πλευρά οικονομική ε, στήριξη και από πλευρά εντολή. Γιατί μα είπε ο Επίτροπο Έντιγκερ προηγουμένω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκή ψηφιακή προσέγγιση και όραμα χωρίς ε, να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ασφάλειας και ότι ενδεχομένως αυτό να είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι η ιδέα ενό ευρωπαϊκού υπολογιστικού νεφου είναι ιδιαίτερα ελκυστική και για εταιρείε όπω η Microsoft και ότι βλέπουμε ότι παίρνουμε πιο σοβαρά πλέον την ασφάλεια στην κυβερνοχώρα, ενδεχομένω πιο σοβαρά από τι άλλα τμήματα του κόσμου. Ευχαριστώ από πλευρά Σοσιαλιστών, η κυρία Καϊλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας ενημερώσατε ε, για τα όσα πράτετε. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ορισμένα στοιχεία Πρόσφατα είχαμε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, διαρροών από αξιωματούχους, για παράδειγμα και συζητήσεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όλα αυτά οδήγησαν και σε πολιτικές εξελίξεις. Θα ήθελα να μου πείτε εάν και οι πολιτικοί μπορούν να συμβάλλουν ε, και αν μπορεί να υπάρξει προστασία και των πολιτικών για, και πώς μπορεί αυτό να στηριχθεί οικονομικά, γιατί δάλλως ε, πώς μπορούν και οι ίδιοι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια. Θεωρείτε ότι μπορείτε ε, να δώσετε μια τέτοια υπηρεσία και εσείς αλλά και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλήσετε και για την κρυπτογράφηση και πόσο σημαντική είναι. Θα ήθελα να μας πείτε για ορισμένες εφαρμογές που έχουν κρυπτογραφική πρόσφατα όπως είναι το Viber και το WhatsApp. Νομίζετε ότι αυτό είναι ασφαλές ή ότι μόνο με τη χρήση αυτής της ε, μιας συσκευή μπορεί να διαρρεύσει το περιεχόμενο. Επίσης για το blockchain θα ήθελα να ρωτήσω γιατί έχουμε το αντίθετο. Οι τρομοκράτες και οι εγκληματίε ε, εποφελούνται των νέων τεχνολογιών. Πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βρούμε την ισορροπία και του ελέγχου αλλά και της μη παρεμπόδισης των νέων τεχνολογιών. Γιατί λέτε ότι γνωρίζουν τα καταστήματα τι θέλουμε να αγοράσουμε και μας κάνουν προτάσεις. Μπορούν ακόμα και να εντοπίσουν τη διάθεσή μας, αν έχουμε προβλήματα υγείας, βάσει των αναζητήσεων που κάνουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια στην κυβερνοχώρο και πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν εάν θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση του προπολογισμού, γιατί υπάρχουν τρομοκρατικέ ενέργειε, όλοι αυξάνουν τον προπολογισμό του για την ασφάλεια και εμεί τον μειώνουμε. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένε προτάσει, τι οποίε θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, e Ευχαριστώ. Από πλευρά e Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρούμε το ρόλο του ΕΝΙΣΑ πολύ σημαντικό για τα θέματα της προστασίας της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Γι' αυτό και όταν η Ελλάδα ζήτησε να πάρει την έδρα του ΕΝΙΣΑ στο Ηράκλειο της Κρήτης, δεν το έκανε τυχαία, διότι ζήτησε να εγκατασταθεί στο χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ένας χώρος στον οποίο αναπτύσσεται η έρευνα και των δικτύων, ένας χώρος στον οποίο αναπτύχθηκε η Forthnet, μια μικρή εταιρεία η οποία όμως σήμερα είναι μια μεγάλη εταιρεία τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Ένας χώρος που είναι ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης που έχει εξειδίκευση στα θέματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ως βουλευτής του Ηρακλείου της Κρήτης το 2012 και 2013 αντιμετώπισα τις μεθοδεύσεις της ηγεσία του ΕΝΙΣΑ ο οποίος ήθελε να φύγει από το Ηράκλειο πιέζοντας να πάει στην Αθήνα και σε δεύτερη φάση να φύγει εκτός Ελλάδος, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το επιχείρημα που είχαν, γιατί ασχολήθηκα στενά με το θέμα, ήταν η δίθεν άσχημη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει θεραπευτεί μετά από πολλές παρεμβάσεις δικές μου και άλλων βουλευτών. Αλλά βλέπω λοιπόν μια προσπάθεια να φύγει ο Ενίσα, την οποία μεθοδεύει η ηγεσία, του Ενίσα και πέτυχε να σπάσει ο Ενίσα σε δύο κομμάτια κύριε Πρόεδρε. Σε ένα χώρο που θα είναι διοικητικό κέντρο και θα παραμείνει στο Ηράκλειο και σε ένα επιχειρησιακό κέντρο στην Αθήνα που σημαίνει διπλά έξοδα, που σημαίνει μεταφορές υπαλλήλων, που σημαίνει λειτουργίες τέτοιες. Ενώ στο Ηράκλειο έχετε 4.500 χώρο για να υπάρξει η λειτουργία και ταυτόχρονα μεθοδεύεται μια κατάσταση και λέτε, και το λέει και η Επιτροπή εδώ προϋπολογισμού, στην οποία μεθοδεύσατε να πάρθει μια απόφαση. Τι λέει λοιπόν, ότι το ενίκιο στην Αθήνα δεν πληρώνεται, διότι η ελληνική κυβέρνηση προφανώς είχε οικονομικά προβλήματα. Να μείνετε στο Ηράκλειο, όπου εκεί υπάρχει η λύση και όχι να δημιουργείτε το πρόβλημα. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει το πρόβλημα των επιπλέον εξόδων και όχι η ελληνική κυβέρνηση. Και δεύτερον, ακούστε επιχείρημα γιατί θέλουν να πάνε στην Αθήνα όπου δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σχολείο. Όπου εκεί πληρώνονται ιδιωτικά σχολεία για να υπάρχουν. Λέει λοιπόν στο Euroactive Employees of the agency complain about schools and sparse job prospects. Και ε, αυτό την πυροβολή της ε, προοπτικές εργασίες για τους τοπικούς εργαζόμενους. Φίλοι σας, ήρθατε για να δουλέψετε. Να καταλάβετε λοιπόν ότι οι μεθοδεύσεις σας δεν περνάνε. Πέρυσι σας είπα τα ίδια και μην γελάτε κύριε. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ είναι Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είστε ελεγχόμενος. Δεν θα μας κάνετε έλεγχο εσείς. Καταλάβατε. Να συμπεριφέρεστε σωστά σε αυτούς που έχουν εκλεγεί ως Ευρωβουλευτές και να μην χαμογελάτε. Και να μην χαμογελάτε. Κύριε Πρόεδρε, θα τον ανακαλύψετε στην τάξη. Να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Να τον ανακαλέσετε στην τάξη. You have to tell this Θα πρέπει να πείτε σε αυτόν τον κύριο να μην χαλμογελάει και να ακούει τους ευρωβουλευτές με όλο το σεβασμό που αρμόζει. Δεν δέχομαι τον τρόπο με τον οποίο μας φέρετε. Ήρθατε εδώ όχι για να χαμογελάτε ηρωνικά, αλλά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ε, ο χρόνος σας ομιλίας έχει τελειώσει πριν από ένα λεπτό. Παρακαλώ, λοιπόν, μείνετε στους κανόνες της Επιτροπής μας. Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, Πρόεδρε, ε, παρακαλώ να, ε, να, να φέρεστε με σεβασμό στους Ευρωβουλευτές. Μάλιστα, έχουμε πλήρη. Όχι, δεν με σέβετε. Εσείς δεν σέβεστε όλους μας, διότι δεν κλείνετε την ομιλία σα που έπρεπε να έχει τελειώσει πριν από ένα λεπτό. Ωραία, οπότε με σταματάτε εμένα, έτσι κύριε Πρόεδρε. Μα δεν τελείωσα. Οι υπόλοιποι μίλησαν για δυόμιση λεπτά. Δεν τελείωσε ο χρόνος μου. Okay. Uh, If I may, please, Madam, Madam Callas, to take a Παρακαλώ κύριε Κάλλας, έχετε τώρα το λόγο εξ ονόματος της Άλντε. Okay. Well, it was not really clear what was the problem here, but... Δεν κατάλαβα καλά ποιο ήταν το πρόβλημα, αλλά παρακα... εγώ θα επανέλθω στα θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου. Um, so, um, about the cybersecurity issues, I, I totally agree with you that... Uh, εγώ θεωρώ ότι τα όσα είπατε για την ιδιωτικότητα των στοιχείων ε, και τους κανόνες προστασία των στοιχείων θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι το ίντερνετ δεν ε, σχεδιάστηκε για τους λόγους για τους οποίους το χρησιμοποιούμε τώρα, οπότε υπάρχουν θέματα ασφάλειας πολύ σοβαρά και αν και έχουμε συζητήσει πολύ για τις κυβερνήσεις, το ρόλο τους και το ρόλο των θεσμών και διάφορα άλλα στοιχεία της αλυσίδας, της αλυσίδας που είναι ο κόσμος και οι εταιρείε. πιστεύω ότι από την πλευρά των κυβερνήσεων οι κυβερνήσεις έχουν κάνει πολλά ώστε να ανασφαλίσει οι επικοινωνίες τους και οι υπηρεσίες πιο ασφαλείς, αλλά αδύναμος, η αδύναμη κρίκη είναι οι άνθρωποι και οι εταιρείε που δεν ε, ενημερώνουν πάντα το λογισμικό τους και δεν κάνουν τα απαραίτητα βήματα ώστε να ε, έχουν αρκετή ασφάλεια. Το ερώτημά μου λοιπόν σχετίζεται με όλα αυτά. Πώς βλέπετε τον ρόλο ή την χρήση των ε, κρυπτογραφημένων ταυτοτήτων. Γιατί πολλά προβλήματα για τον κόσμο προκύπτει από την κλοπή ταυτοτήτων στο ίντερνετ και μετά την ε, διάπραξη διαφόρων ε, δικημάτων ε, μπορεί κάπως να γίνει ώστε ε, ο κάθε άνθρωπος να πρέπει να έχει δικό του κωδικό, θα είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιεί κανείς τις επικοινωνικές υπηρεσίες με πιο ασφαλή τρόπο και να μειώνονται έτσι κίνδυνοι. Ποια είναι η άποψή σας επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα πάμε στον επόμενο, στο επόμενο μιλητή που είναι ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω για μας όλους έχει σημασία η Ενίσσα να συνεχίσει στο μέλλον και να επεκτείνει τις δραστηριότητε για την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο και κατανοώ τον εκνευρισμό ορισμένων εδώ που δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια ε, στον κυβερνό χώρο αλλά το αντίθετο, το χάος και η καταστροφή. Δεν είναι όμως δική μας υπόθεση αυτή. Έχουμε δύο μπλοκ, ε, την ιδιωτική ζωή και τη διαφάνεια που μπορεί να συγκρούονται έχει σημασία η ιδιωτική ζωή να έχει τη δυνατότητα να κάνει ασφαλείς επικοινωνίες. Εντάξει, η κρυπτογράφηση είναι πολύ σημαντικό και το blockchain επίσης και η επιστημονική υπηρεσία του Κοινοβουλίου, η ΣΤΟΑ, πρόσφατα έκανε μια διάσκεψη, ένα σεμινάριο για τις κβαντικές τεχνολογίες. Ε, τι γίνεται με τις ασφαλείς επικοινωνίες που δεν μπορούν να παραβιάζονται, να υποκλέπτονται, να παρακολουθούνται. Ε, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για ασφαλή ζωή στο μέλλον. Ε, απόλυτα ασφαλείς λοιπόν συνδέσεις αποτελούν τη βάση για ένα σταθερό πλαίσιο και με ενδιαφέρει ε, το πώς δραστηριοποιείται και ο Νίσα. Ευχαριστώ. Next speaker, η σύγχρονη Ευρώπη είναι ψηφιακή, άρα χρειαζόμαστε περισσότερα μέτρα ασφαλείας για να βελτιώσουμε την ε, ε, δυνατότητα λειτουργίας του ΕΝΙΣΑ και να υπάρχει και μια ισχυρή εντολή αν θέλουμε να έχουμε και αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρώτα απ' όλα ως Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα θα πρέπει να υποστηρίξουμε την οδηγία για την εφαρμογή της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο γιατί αυτό είναι το υπόβαθρο. Δεύτερον, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον ΕΝΙΣΑ για να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στα πλαίσια του Horizon 2020 με τα ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα και να υπάρχει πρόσβαση σε πολλά ε, έργα σε αυτή την ε, υπόθεση αυτό το κλάδο. Υπάρχουν πολλές συστάσεις επίσης του ΕΝΗΣΑ σε διάφορες εκθέσεις προς τη βιομηχανία, προς τα νοσοκομεία ας πούμε. Πριν από λίγο καιρό εκδώσατε και έχει μεγάλη σημασία να εφαρμοστούν αυτές οι συστάσεις διότι τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου υφίστανται οι συστάσεις, καταναούμε το πρόβλημα και τώρα πρέπει από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε και να τα εφαρμόσουν οι ενδιαφερόμενοι. Και το τελευταίο έχει να κάνει για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ασφαλείας στην Ευρώπη και του κλάδου αυτού. Έχει έρθει η ώρα να ε, επενδύσουμε και εκεί και ο Ενίσα είναι πολύ καλή πηγή πληροφοριών, γνώσης και υποστήριξης ε, Υπάρχει τώρα ένας ολόκληρος κλάδος ασφάλειας, security by design, όπως και privacy by design. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Χέρμπρεχτ, καλώ ορίσατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω μαζί με άλλους συναδέλφους. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και εμείς ξέρουμε να το εκτιμούμε. Πραγματικά προσπαθείτε να ε, αναπτυχθείτε και προς την κατεύθυνση που επιθυμούμε εμείς. Έχω δύο ερωτήσεις, γιατί δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δραστηριότητες σας όσο άλλοι συνάδελφοι. Πώς συνεργάζεστε με ε, άλλους φορείς, με την Ευρωπόλα ας πούμε, συνεργάζεστε πιο πολύ με τη Frontex, ε, τι κάνετε εκεί σε αυτό το τομέα για θέματα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού που μας ενδιαφέρουν ε, και την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια ε, ψηφίσαμε την οδηγία και το βασικό κανονισμό για τα ε, δεδομένα για μεγαλύτερη και αστυνομική συνεργασία. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στη δική σας δουλειά επιτόπου και πάρα πολύ συγκεκριμένα. και στην προηγούμενη ομάδα 29 τη λεγόμενη συνεργάζεστε, συμμετέχετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ενδιαφέρει να δω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much, thank you. First of... Ευχαριστώ πολύ κύριε Νάτι. Ευχαριστώ. Στη φινλανδική εκδοχή του σχεδίου μερίσης διάταξης λέει ανταλλαγή απόψεων για την ψηφιακή βιομηχανική πρωτοκαθεδρία, ενώ στα αγγλικά λέει μόνο ε, ευκαιρία. Οπότε είναι πρωτοκαθεδρία αυτό ή, ευκαιρία. Βοηθάει ο Ενίζα να είμαστε πρωτοπόροι ε, στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή και στην ψηφιοποίηση. Ήταν πολύ σημαντικό γιατί το συζητήσαμε αυτό στην ψηφιακή ενιαία αγορά ότι εξαρτώμαστε πάρα πολύ από υπηρεσίες ασφαλείας άλλων ε, ε, υπήρων. Ακούσαμε και τι γίνεται στη Φιλανδία, τι γίνεται στην Ευρώπη, αλλά ε, ε πολλές χώρες, εταιρείες, βιομηχανία μπορεί να επαφίονται σε ρωσικά συστήματα, ασιατικά ή αμερικανικά. Μήπως πρέπει να έχουμε και εμείς κάποια στρατηγική για να έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες, ικανότητες κτλ και εγώ εκεί το εντάσσω στη ψηφιακή βιομηχανία γιατί είναι μεγάλες εταιρείες που χρειάζονται πολλά στοιχεία από δορυφόρους, πολλούς υπολογιστέ, νέφη κλπ. Έχουμε λοιπόν καμιά στρατηγική. Ο Ενίσσα βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Συνεργάζεται. Γιατί αυτά λένε στην ημερήσια διάταξη στο σημείο 13 τα φιλανδικά και είναι ένας παράγων ανταγωνιστικός στην Ευρώπη. Είμαστε σε καλύτερη μοίρα για την ασφάλεια από άλλους. Το έχω πει επανειλημμένα. Ε, εγώ έχω ένα πολιτικό όραμα, άλλοι έχουν τις γνώσεις όμως και θέλω να με διαφωτίσουν. Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση μόνο, συμπληρωματική μετά από την εκνευρισμένη παρουσίαση ε, του συναδέλφου, συνήθως ε, χειριζόμαστε διαφορετικά τους προσκεκλημένους. Μη αποκομίστε λάθος εντύπωση. Ξέρω ότι το θέμα αυτό μας απασχολεί εδώ και καιρό και το θέμα της έδρας ήταν ιδιαίτερο. Δεν το έχω ζήσει με κανένα άλλο οργανισμό αυτό. Και έχει και θέμα ουσίας, έτσι, και πρόβλημα στην ουσία. Και θέλω να επανέλθω σε αυτό, γιατί Θέλω να σας ρωτήσω, γνωρίζω ότι έχετε δυσκολίες να βρείτε ειδικού που χρειάζεστε ε, όσο κανένας άλλος οργανισμός για αυτό το περίπλοκο θέμα. Και αυτοί οι ειδικοί και κυβερνόμονες πρέπει να έρθουν από όλο τον κόσμο. Και ανέκαθεν ήταν πρόβλημα αυτό. Δεν έρχονται και οι ειδικοί. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο οργανισμός αν δεν έχει τους ανθρώπους που χρειάζεται. Και αν είναι πρόβλημα η έδρα, θα πρέπει να τα λέμε και να μπορούμε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα ανοιχτά, ειλικρινά, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε εχθρικοί απέναντι σε μια χώρα. Δεν πρόκειται καν για μια χώρα. Ε, απλώς θα πρέπει να φύγουμε από ε, ένα ε, τόπο που είναι σε ένα χαζό νησί, λέει ο μιλητής. Ε, αυτά έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και συνέπειες. Πρέπει να έχετε τους καλύτερους εμπειρογνώμονες. Αλλιώς όσο καλός και έναν οργανισμός δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Έχετε ακόμα δυσκολίες λειτουργικές ή βρίσκετε εμπειρογνώμονες που να θέλουν να έρθουν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. I don't see any. I would like to ask uh, European Commission uh, for... Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σχόλια. Ο κύριος Πολ Τιμέρς. Από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Διευθυντής, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για τη δυνατότητα που μας δίνετε να πούμε δύο λόγια, ακριβώς στο πλαίσιο της ε, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ε, και πώς αυτή αποτελεί οικονομική δυνατότητα και υπό το φως και του νέου πακέτου ε, που δημοσιεύθηκε πριν από δύο ημέρες. Έχουμε, ας πούμε, και το σχέδιο δράσης για το ζήτημα αυτό, ακριβώς με τη δημόσια διοίκηση και την ασφάλεια στη δημόσια διοίκηση στην ηλεκτρονική και πώς ακριβώς μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και για ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές υπογραφές και το καθεξής. Και το Κοινοβούλιο όσο έχει ε, υπερψηφίσει ένα ψήφισμα το οποίο είναι ένα από τα πιο επιτυχή αποτελέσματα ε, σωστής συνεργασίας και αποστέλνει το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική ταυτοποίηση το χρησιμοποιούμε και στη δημόσια διοίκηση και στον εμπορικό χώρο. Είναι ένα τομέα όπου η ΕΝΙΣΑ μα έχει δώσει ε, πολλέ συμβουλέ ακριβώ για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στον κανονισμό. Και το ε, σχέδιο δράση για την ελληνική Διακυβέρνηση εκεί βασίζεται. Τώρα στο πακέτο υπάρχουν και άλλα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την τυποποίηση και εκεί η ασφάλεια των γυμνοχώρων είναι κέριο ζήτημα. Ένα στοιχείο εκεί είναι ότι θα θέλαμε να έχουμε την ασφάλεια του σχεδιασμού by design, όντω, Επομένω, αυτοί που χρησιμοποιούν πρότυπα ICT, ε, τεχνολογία τη πληροφορία, θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ασφάλεια του κυβερνοχώρα από την αρχή και να παραπέμπουμε και σε πρότυπα. Θα γίνει αυτό. Θα μιλήσουμε και για την τυποποίηση στην ασφάλεια του κυβερνοχώρο για αναδυόμενου κλάδου όπω είναι το υπολογιστικό νεύχο και το διαδίκτυο των αντικειμένων και να δούμε ε, τι, τι οδηγία θα υιοθετηθεί ακριβώς και για αυτό το ζήτημα και εκεί ο ΕΝΗΣ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Επανέρχομαι στην οικονομική δυνατότητα. Ε, μιλούμε πολύ για απειλέ. Για παράδειγμα, αυτή την εβδομάδα ασχολούμαστε με τα νοσοκομεία που ε, τους, ε, προσπαθούν να τους εκβιάσουν ε, για λίτρα, χρηματικά ποσά. Συνεχώ ακούμε απειλέ εδώ, απειλέ από εκεί. Όμω υπάρχουν και οικονομικέ δυνατότητε. Γιατί αυξάνεται κατά 7,5% η αγορά κάθε χρόνο. Και η Ευρώπη έχει μια πολύ καλή φήμη. Είμαστε αξιόπιστοι, έχουμε επιχειρήσει ε, που προσελκύουν μεγάλο ενδιαφέρον και από ξένο κεφάλαιο, αλλά εξαιτία τη τεχνογνωσία είμαστε πολύ ελκυστικοί. Έχουμε εξαιρετικέ δυνατότητε δικτύωση ε, και ασφάλεια. Επομένω, υπάρχει μια βάση, αλλά θέλουμε να κάνουμε και περισσότερα. Θέλουμε να υπάρξει μία ε, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να ενισχύσουμε την ε, εικονότητα στην Ευρώπη και έναν αριθμό συνοδευτικών μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος πιστοποίησης στην Ευρώπη. Ένα είδος ε, εμπορικού σήματος, ε, ότι δηλαδή η Ευρώπη είναι ο πιο ασφαλής η πιο ασφαλή περιοχή ω προ την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, κάτι τέτοιο τέλο πάντων, ένα σήμα που να μα δείχνει ε, ω του πιο ασφαλεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Διευθυντά, αν θέλετε κι εσείς ε, να απαντήσετε και να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω στα γερμανικά, ε, γιατί στη μετρική του γλώσσα κανεί μπορεί να εκφράζεται καλύτερα, να παίρνει καλύτερα το μήνυμα. Αρχίζω από την έδρα για να ε, ξεφύγει αυτό το συναισθηματικό θέμα, να το διεκπαιρεώσουμε στην αρχή και να προχωρήσουμε. Κρίμα που αποχώρησε ο συνάδελφος. Πραγματικά θα τον προσκαλούσα, το έχω κάνει επανειλημμένα, να έρθει επί τόπου και να δει πώς έχει κατάσταση. Γιατί πολλά γράφει και ιδιαίτερα ελληνικός τύπος που τότε δεν ισχύουν. Ε, και θέλω να το πω και αυτό. Να σας πω μερικά στοιχεία, δεδομένα αντικειμενικά πρώτον. Από το 2013 έχουμε δύο έδρες με τον νέο κανονισμό. Εκεί λέγει ότι η διοίκηση είναι στο Ηράκλειο και τα λειτουργικά επιχειρησιακά είναι στην Αθήνα. Στο μεταξύ έχουμε 94 θέσεις, 94 στο οργανόγραμμα ενίσα, εκ των οποίων 60-65 στο μεταξύ είναι στην Αθήνα. Δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων εδρεύει στην Αθήνα. Και από την Αθήνα λειτουργούμε. Ευχαριστούμε και την ελληνική κυβέρνηση διότι μας ε, διέθεσε το κτίριο ε, και πληρώνει και το νίκη, νίκηση διότι και όποιος θέλει να μας δει ε, είναι πρόσδεκτος ανά πάσα στιγμή, είναι σε ένα καταπληκτικό σημείο και όποιος ζει στην Ελλάδα εδώ και καιρό στα βόρεια προάστια είναι πολύ καλή η ε, ε, δουλειά κοντά μας είναι ο Κοσμοτέ, η Microsoft και τα λοιπά και ε, ό,τι μας χρειάζεται. Εμείς δεν είμαστε ερευνητικό ίδρυμα. Γι' αυτό δεν χωράει η σύγκριση που έγινε με το Force θέλουμε να έχουμε έργα στην Ευρώπη, project στα κράτη-μέλη, να υποστηρίζουμε τις αρχές, τις κυβερνήσεις, ε, την οικονομία. 600.000 το χρόνο έχουμε δαπάνες ταξιδιωτικές για τους ε, υπαλλήλους. Πηγαίνουμε στους πελάτες μας, στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες, στα project, στα έργα τα διάφορα. Και θέλω να πω και το εξής εδώ. Έχουμε ένα άδειο κτίριο το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ηράκλειο, που μας το έχουν τάξει οι τοπικές αρχές. Και στο μεταξύ έχουν επενδυθεί και 14 εκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και είναι μη τελές ακόμα το κτίριο. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν μιλάει κάποιος για ένα σχολείο, καλό είναι να το επισκέφτεται, όχι απλώς να μιλάει γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά και στα αγγλικά. Θα τα συνεχίσω. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, ε, κυρία Νίμπλε, για την στήριξή σας. Θα διατρέξω τα σχόλιά σας και θα απαντήσω με τη σειρά. Σωστά είπε ο κύριος Σέιλερ ότι έχουμε τη βιομηχανία, δημιουργούμε νέες θέσεις απασχόλησης, νέα πρότυπα, πρέπει να προστατευτεί ο ίδιος ο κλάδος. Αυτή είναι η πρόκληση. Βελτιωνόμαστε με τον καιρό και στη Γερμανία με, τις, με τους σχετικούς νόμους ε, ασφάλειας στην τεχνολογία της πληροφορίας κλπ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για την βελτίωσή μας και βελτιωνόμαστε, αλλά ακόμα πολλά μένουν ακόμα να γίνουν. Η τυποποίηση λοιπόν είναι το ένα. Ε, είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και βελτιωνόμαστε, όμως αποτελεί πρόκληση γιατί εργάζονται πολλοί σε αυτόν τον ε, τομέα πολλούς επιμέρους οργανισμούς και εδώ και στις ΗΠΑ Υπάρχει λοιπόν ένας κατακαιρματισμός. Και για να σας δώσω ένα θετικό παράδειγμα, έχουμε τομέα που υπάρχουν ε, κοινά ε, κριτήρια τυπο... αυτοπίσεις τυποποίησης. Η πρόκληση λοιπόν είναι το είπε και ο κύριος Τίμες. Θέλουμε να κάνουμε πολλά. Αλλά για να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η τυποποίηση είναι κάτι το δύσκολο. Και ίσως και με τέτοιες πρωτοβουλίες της Κομισιόν μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια στρατηγική τυποποίηση και εκεί να καταβάλουμε τις προσπαθίες μας. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ε, αμερικανικές επιχειρήσεις ε, προηγούνται, ενώ εμείς καθόμαστε ακόμα και συζητούμε τις ε, λεπτομέρειες. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά είναι πρόκληση. Ε, ελπίζω να σας απάντησα. Μετά για την κρυπτογράφηση που ανέφερε η κυρία Καηλή και άλλοι. Η σημερινή πρόκληση λοιπόν είναι ότι υπάρχουν πολλές τεχνολογίες. Υπάρχει κρυπτογράφηση, υπάρχει πιστοποίηση, υπάρχουν προϊόντα και εργαλεία. Το πρόβλημα μας είναι πώς όλα αυτά θα μπουν στην αγορά. Και τέτοια προϊόντα συνήθως δεν είναι εύχριστα για τον ίδιο τον καταναλωτή τον ίδιο το χρήστη. Επομένω, η ίδια βιομηχανία θα πρέπει να μας δώσει πιο εύκολα και εύχρηστα ε, τέτοια προϊόντα. Δεν... Ε, αν ήταν κάτι πιο εύκολο, δηλαδή απλά πατούσε κάποιο ένα κουμπί στο email του και γινόταν η κρυπτογράφηση, τότε θα το χρησιμοποιούσε ο καθένα. Αλλά δεν ε, συμβαίνει αυτό προ το παρόν. Αν δείτε για τι ηλεκτρονικέ ταυτότητε. Έχουμε στην Ευρώπη ηλεκτρονικέ ταυτότητε με κάρτε. Στη Γερμανία έχουμε τέτοιε ταυτότητε και στο Βέλγιο και στην Αυστρία και στην Εστονία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πάντα συμβατά όλα αυτά μεταξύ του και κάποιε φορέ είναι και ακριβά. Ω Γερμανό υπήκο μπορώ να σα πω ότι έχουμε ηλεκτρονικό διαβατήριο που πραγματικά είναι εξαιρετικά ασφαλέ, όμω χρειάζεται κανεί ένα, ε, ε, ένα ειδικό ε, μηχάνημα ανάγνωση αυτή τη κάρτα ε, χρειάζεται το, το λογισμικό και μετά υπάρχει το πρόβλημα ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλοί χρήστε, δεν αναπτύσσονται και αντίστοιχε εφαρμογέ. Υπάρχουν λοιπόν οι ευκαιρίε, αλλά χρειαζόμαστε πιο εύχρηστα προϊόντα, πιο απλά στη χρήση του. Μίλησα για τη σχετική οδηγία. Εμείς λοιπόν από τον ΕΝΙΣΑ προσπαθούμε να τα στηρίξουμε όλα αυτά. Είχαμε και τον σχετικό μήνα για την ασφάλεια στην κυβερνοχώρο που συνεργαστήκαμε και με τα κράτη-μέλη. Αλλά εκεί χρειαζόμαστε και πολλούς πόρους. Πώς συνεργαζόμαστε λοιπόν με ε, τον κλάδο και τους οργανισμούς. Να σας δώσω ορισμένα ονόματα. Για τους οργανισμούς ε, συνεργαζόμαστε στενά με την Μπέρεκ, με τον Ιουλίζα. Λίζα. Έχουμε πολύ τακτικά συναντήσεις με τους επιμέρους φορείς, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχει λοιπόν ένα δίκτυο διαλόγου. Κάποιος ανέφερε τη Frontex. Εμείς δεν συνεργαζόμαστε με τη Frontex. Γιατί νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κοινό πεδίο αρμοδιοτήτων. Όμως ε, όπου υπάρχει IT στην εντολή άλλων οργανισμών συνεργαζόμαστε και όπου αυτά συνδέονται με τη βιομηχανία προσπαθούμε να τα συμπληρώσουμε. Αν δείτε με την Κομισιόν, το πρόβλημα είναι ότι με την Κομισιόν, η Κομισιόν δεν μπορεί να συνομιλήσει με 50% επιχειρήσει. Προσπαθούμε λοιπόν από τον ΕΝΙΖΑ να διοργανώνουμε εκδηλώσεις ε, και να έχουμε εκδηλώσεις ε, και δικτύωσης με τον κλάδο και ανέφερε Φιλανδή συνάδελφο ε, πώ μπορούμε να συνεργαστούμε με την f που είναι μια φιλανδική ε, εταιρεία. Δημιουργούμε λοιπόν ένα δίκτυο και πριν από μερικές εβδομάδες εξετάσαμε το τι συμβαίνει και στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας και των πληρωμών και πώς μπορεί εκεί να υπάρξει ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Επομένω, έχουμε ένα δίκτυο διαλόγου συζητήσεων, συστάσεων και μετά κλαδικά προσπαθούμε ε, να εξετάσουμε κάποια πολιτικά προγράμματα. Είμαστε μικρός οργανισμός, επομένω η πρόκληση είναι ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε ορισμένες μόνο προτεραιότητες και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε στη νέα εντολή. 84 οργανικές θέσεις ανέφερα. Από αυτές τις 84, μόλις 48 είναι ε, προσωρινή υπάλληλη, temporary. Γι' αυτό το θετικό είναι ότι μπορούμε να λάβουμε πόρους από το εθνικό πλαίσιο, αλλά μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξετάσουμε ποια θα είναι η στρατηγική του ΕΝΙΣΑ. Αναφέρθηκε το ζήτημα των ε, προσλήψεων. Ε, είναι καλύτερα από τότε που πήγαμε στην Αθήνα αλλά υπάρχει άλλη πρόκληση, γιατί αν δείτε ε, την κατάσταση στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχουμε στη Βόρεια Ευρώπη ανάπτυξη οικονομική, επομένως οι Γερμανοί και οι Σουηδοί δεν θέλουν ιδιαίτερως να πάνε στην Αθήνα. Επομένω, δυσκολευόμαστε να προσλάβουμε ε, ανθρώπους με ψηλές δεξιότητες, αλλά είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει τόσο οικονομική, μεγάλη οικονομική διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου. Και αυτό είναι ζήτημα. Ελπίζω να απάντησα. Αν έχω ξεχάσει κάτι, θυμίστε το μου. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι απαντήσατε στα περισσότερα από τα ερωτήματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας και για όλε τις δραστηριότητε του ΕΝΙΣΑ. Βλέπετε ότι και εμεί κατανοούμε τη σημασία ε, της ασφάλειας στην κυβερνοχώρο, αλλά και της ε, παροχής ορισμένων οικονομικών ε, δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θεσμολό Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο επόμενο θέμα παρουσίαση της εκθέσης Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινοτομίας και Τεχνολογίας. European Institute uh, Innovation and Technology, and we've got a presentation of the of Παρουσίαση έλεγα της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ενεκτικού Συνεδρίου και θέλω να σας θυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο μόλις έκανε μια μελέτη και έκθεση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τη συμμόρφωσή του. Ο κύριος Άλεξ Μπρένιγκ Μέιερ είναι παρόν για να μας παρουσιάσει ε, στην Επιτροπή μας δηλαδή τα πορίσματα της έκθεσης αυτής ε, στο βαθμό που είναι δική μας αρμοδιότητα. Επίσης ε, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον Επίτροπο κύριο Τίμπορ Ναύρασιτς στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας και πώς Καπάει και τις επιδόσεις του. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή μετά τον Επίτροπο. Να ακούσουμε τις απόψεις του Ελεκτικού Συνεδρίου. Έχετε το λόγο, παρακαλώ, και καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ήτρε. Είμαι πολύ πολύ ε, ικανοποιημένος από την οπτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε μία από τις ειδικέ μας εκθέσεις που εστιάζει στην απόδοση ε, μιας σημαντικής ε, υπηρεσίας της CIT που εδράζει στην Βουδαπέστη. Αυτός ο έλεγχος δεν, δεν ελέγχει τα οικονομικά και τη συμμόρφωση, αλλά την αποτελεσματικότητα της επένδυσης της Ευρώπης αυτή στο EIT. Εγώ είμαι αναφέρον μέρος, μέλος του Συμβουλίου του Ελληνικού Συνεδρίου ε, και πολύ ευτυχής είμαι που έχουμε αυτή την επαφή με την Επιτροπή σας. Επίσης έχουμε υποβάλει αυτή την έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και ε, εκεί αφορούσε την, τα οικονομικά, ενώ τώρα το περιεχόμενο, την ουσία. Επίσης να τονίσω το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα θέματα. Η EIT είναι τμήμα του, του οργανογράμματος της Κομισιόν και η ΕΑΚ e είναι υπεύθυνη, η e RTD είναι επίσης υπεύθυνη για τμήματα που αφορούν την έρευνα και την κοινοτομία. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία του RTB για την εγκαθίδρυση ενός ε, Συμβουλίου ε, καινοτομία απαιτεί την προσοχή από δική σας πλευράς. Άλλο σημείο ε, για τα επικεφαλίδες και με χαρά θα απαντήσω στις παρατηρήσεις σας Το EIT στη Βουδαπέστη στοχεύει και εστιάζει στην καινοτομία και την ανάδειξη και την προώθηση αυτής γιατί η καινοτομία είναι αδύναμη στην Ευρώπη. Αυτό που κάνουμε είναι ε, να ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και να τις βοηθήσουμε σε αυτό που αποκαλείται τα ε, κέντρα και ε, γνώσης καινοτομία, τα KICS, που είναι πολύ σημαντικά για τις ε, για βιομηχανίες. Έχουμε επισκεφθεί τρεις για την ενέργεια, για το περιβάλλον. Έχουμε ενοποιημένους ε, εταίρους και εδώ ε, μας είπε το ΙΑΙΤ e ότι έχουμε ήδη 800 συνεργάτες. Η ευρωπαϊκή λοιπόν συνεργασία και καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε επισκεφτεί δε διάφορα κέντρα γνώσης ε, τέτοιου τύπου και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν εντωμεταξύ εντυπωσιακέ πρωτοβουλίε για πρωτοβουλίε και υπάρχει και μεταφορά από την έρευνα. προς τις startup. Κάτι άλλο είναι ότι ακούμε, πρέπει να ακούσουμε πολύ προσεκτικά τι συμβαίνει επί τόπου. Ελέγχοντας τα κίξ αυτά τα ναι, τα, τα αυτά τα, κέντρα, ε, νομίζω ότι διαπιστώσαμε ότι ετησίω πρέπει να εκπονήσουμε χίλιε σελίδε για μια εφαρμογή ετήσια. Και αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και έπειτα είναι ετήσια αν και ε, τα δικό μας ε, προγράμματα ε, διαρκούν πολύ περισσότερο από ένα χρόνο. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον των προγραμμάτων αυτών και δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό βοηθά για την καινοτομία. Να υπάρχει δηλαδή τόσο λίγη βεβαιότητα για το μέλλον. Μια άλλη παρατήρηση Κάτι που μας είπε ένας εταίρος στο πρόγραμμα είναι ότι ε, διαπιστώνει τόσο πολλά προβλήματα σε αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ δύσκολο να ε, δυσδύσουμε και μας πήρε πολύ η προσπάθεια να το δεχτούν και να συνεργαστούν. Ευτυχώς το καταφέραμε. Αλλά βλέπετε ότι το γραφειοκρατικό ε, ο γραφειοκρατικός φόρτος είναι μεγάλος και από τη μια πλευρά τα προγράμματα ε, που έχει εφεύρει το ΙΕΤΗ μέσα στην ε, πλαίσιο της αποστολής και σε σχέση με τα πανεπιστήμια, τις επιχειρήσεις και τα ερευνητικά κέντρα ίσως να μην υπάρχει πάντοτε μια εξαιρετική, εξαιρετικός συντονισμός η χρηστή λειτουργία του ΙΕΤΗ στην Βουδαπέστη εν γέννη ε, παρεμποδίζεται από, από περίπλοκο λειτουργικό πλαίσιο, επιχειρησιακό πλαίσιο και σοβαρά προβλήματα διαχείρισης. Έχουμε καταλήξει σε κάποιες συστάσεις ε, και θα τις αναφέρω συντομία. Η πρώτη, το πρώτο θέμα θα πρέπει να είναι η νομική βάση του EIT, η αναθεώρηση δηλαδή του συστήματος χρηματοδότησης και για παράδειγμα ο αποκλεισμό συμπληρωματικών δραστηριοτήτων διότι δεν προκύπτουν και άρα δεν είναι ένα αποτελεσματικό τμήμα του μοντέλου. Η EIT θα πρέπει να επεκτείνει τις συμφωνίες ε, ε, χωρί για υποτροφίες ε, δίνοντας ε, τις στα κέντρα γνώσεων και θα πρέπει να συνάψει αυτές τις συμφωνίες ε, υποτροφιών νωρίτερα ώστε να είναι να επικρατεί νομική βεβαιότητα από την πρώτη μέρα του χρόνου και αυτό πρέπει να, που πρέπει να ξεκινήσουν τα προγράμματα. Η ΑΕΤ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον αντίκτυπο της μόχλευσης και χρειάζεται μεγαλύτερη ε, αυτονομία σε σχέση με την DGEAC. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιεί περισσότερο την ευελιξία που υπάρχει στο ορίζοντας 2020. Ε, οι κανόνες ε, θα πρέπει να είναι πιο προσαρμοσμένοι στις ανάγκες ε, των ε, εταίρων στα κέντρα γνώσης και τέλος θα πρέπει το EIT να επιλύσει τα προβλήματα στελέχωσης δεν έχει το απαραίτητο προσωπικό και η... τα ανώτερα στελέχη ακόμα είναι υπό πρόσληψη και θα πρέπει να βελτιώσει τις αναλύσεις της. Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή και η ΑΕΤ έχουν δεχτεί όλες μας τις συστάσεις και στη διάρκεια του ελέγχου η ΑΕΤ ήδη ξεκίνησε κάποιες από τις κινήσεις που έπρεπε προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι αρκετές, αλλά πάντως προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ο Επίτροπος ε, έχει φτιάξει ένα πάνελ ε, υψηλό επίπεδου για να τον συμβουλεύει για το μέλλον της ΑΕΤ και χτες τον επισκέφθηκα και μου είπε ότι αυτή η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη διότι στηρίζει την περαιτέρω ε, ανάπτυξη του ε ΙΑΙΤ και τη βελτίωση της λειτουργίας του και των κέντρων γνώσης. Κυρίε και κύριοι, αυτή ήταν η σύντομη μου εισήγηση και ευχαρίστως θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας και θα σας δώσω περισσότερες ε, λεπτομέρειες αν ε, το επιθυμείτε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάντα σημαντικές για μας, για την Επιτροπή Ήτρε. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Έλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ του κύριε Μπένιγμαϊρ. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ε, είναι πολύ ενδιαφέρον που αναλαμβάνεται αυτό το είδος το, κομμάτι του διαλόγου με το ελεγκτικό συνέδριο. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι κομμάτι του διαρθρωμένου διαλόγου ανάμεσα στα δύο θεσμούς και είναι αυτός ένας από τους λόγους που διάβασα προσεκτικά αυτή την έκθεση και καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες ε, που εκφράσατε. Η ερώτησή μου ε, αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί. Πιστεύετε πως η πρόκληση μπορεί να είναι η, το πλαίσιο και οι κανόνες που έχουμε επιβάλει στο γιατί είναι το ίδιο, βέβαια είναι ένα, μια μονάδα μόνη της, αλλά ε, παλιότερα συζητήσαμε για το θέμα της απλοποίησης ε, των κανόνων. Είναι συστηματικό το πρόβλημα, συστημικό μάλλον ή προκαλείται από τους κανόνες. Γιατί δεν μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα πρόγραμμα απλοποίησης γιατί οδηγούσε σε πολλές παρεξηγήσεις και προβλήματα για το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα. Δεύτερον, από μια προπτική μεταγενέστερη, τι χρονοδιάγραμμα καλύπτει αυτή η έκθεση. Δηλαδή, στις αρχές έχουμε μια εξέταση από την Κομισιόν, ενώ το EIT σχεδόν ήταν ανύπαρκτο. Δεν ήταν πολύ ε, σκόπιμο αυτό. Και δεύτερον, τώρα το, αυτά που πρέπει να διορθωθούν έρχονται από εσά. Η έκθεσή σας καλύπτει κάποια πρόσφατη περίοδο. Ποια περίοδο καλύπτει. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν θα πρέπει να έχετε την εντύπωση ότι αυτή η σύντομη περίοδος εδώ όπου έχουμε μια ομάδα εργασίας για την EIT και απαραίτητο θα καλέσουμε και σας να συμμετέχετε. Φυσικά το ελεγκτικό συνέδριο και η Επιτροπή δεν είναι ο ένας εναντίον του άλλου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστώ και το ελεκτικό συνέδριο για την έκθεσή του αυτή. Για μας από την αρχή ήταν σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, έχει σχέση με την παιδεία. Και δηλαδή από το πρόγραμμα έρευνας που είχαμε, ε, αυτή η έρευνα και τα αποτελέσματα θα πρέπει να διαδίδουν την έρευνά τους και τα αποτελέσματά τους και να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Όχι στη Φλωρεντία δηλαδή στο αρχείο για να έχουμε τα ωραία αποτελέσματά μας εκεί αρχιοθετημένα, αλλά ε, να πηγαίνουν ε, στα αρμόδια ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστημιακά ε, για να γίνονται αυτές οι νέες ιδέες πράξη, δηλαδή από τις επιστημονικές μελέτες να ξέρουμε ε, τι βοηθάει μια νηπιαγωγό ας πούμε ε, για να εκπαιδεύει τα παιδάκια του νηπιαγωγείου για τη γνώση μέχρι την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που δεν θέλει να μερικάζει στους φοιτητές κάτι που είχε μάθει η ίδια πριν από 40 χρόνια αλλά να είναι στην αιχμή του δόρατος της γνώσης και της καινοτομίας. Και από εκεί και πέρα λοιπόν, ε, αρχίζει ενωμένης από τον υπηαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, τα παιδιά μας να είναι σε επαφή με την τελευταία λέξη της γνώσης και της τεχνολογίας και με την ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να έχει και πρόσβαση. Δηλαδή, στη Φλωρεντία που έχουμε τα έγγραφα, να ξεφύγουμε όμως από εκεί και να πάμε στο ψηφιακό πλαίσιο και να είναι πιο εύκολη ακόμα και η πρόσβαση και στη ΣΤΟΑ που είναι η Επιστημονική Επιτροπή του Κοινοβουλίου που είναι, ΣΤΟΑ σημαίνει Scientific and Technical Option Assessment πώς θα σπάσουν αυτά τα σιλό της γνώσης που είναι σε κάθετη ε, δομή δηλαδή και να γίνουν ε, σωλήνες, εγκάρσιοι, οριζόντιοι που να πηγαίνουν παντού και να ποτίζουν, να μην είναι κλειστά σε ένα κάθετο σιλό, να υπάρχει ε, επικοινωνία και με τα Αυτό βασικά νομίζω είναι η αποστολή του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Πώς υπάρχουν αυτά τα στεγανά και πώς μπορούν να σπάσουν για να έχουμε καλύτερη ε, επικοινωνία. Τι λέγει όλα αυτά το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μούντι. Ευχαριστώ. Από την έκθεσή σας και από τα όσα είπατε σήμερα το πρωί, συμπεραίνω ότι έχετε την εντύπωση ότι τα κέντρα γνώσης και τα EITs κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, επιβεώνω ότι θεωρείτε ότι και πρέπει να επιλύσουμε ζητήματα, αλλά και να δούμε πώς ε, κινούνται προς το παρόν. Με αυτό το σκεπτικό δεν κατανοώ ακριβώς γιατί θέλετε να αναθεωρήσετε τη νομική βάση. Επικρίνετε βεβαίως ε, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, αλλά πώς θα έπρεπε να τότε να τα διορθώσετε αυτά τα προβλήματα και όχι να επανέλθετε στην αιτία που είναι δηλαδή αν θέλετε η απαρχή, η νομοθετική βάση ότι δεν αξιοποιούμε στο έπακρον την ευελιξία του 2020 και έχετε δίκιο, όντω έχουμε την εκτεταμένη οικονομική περίοδο, ενώ εδώ πρόκειται για ένα τομέα με αιτήσιο προγραμματισμό. Τελευταίο σχόλιο. Με τα προβλήματα που έχετε εσείς εντοπίσει Έχετε ορίσει χρονοδιάγραμμα για την εξέβρεση και εφαρμογή λύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι από ό,τι βλέπω. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντένις Κρόλιν, τιμωματάρχης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρένικ Μάιερ και τους αδέλφους του για την έκθεση. Το EIT δεν είναι εδώ, όμως μπορώ να μιλήσω εξ και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του EIT. Το πρώτο που πρέπει να τονίσουμε λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Μπένικ Μάιερ παρουσίασε την έκθεση Μία έκθεση που έχει γίνει αποδεκτή στο σύνολό τη από το EIT και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να το επιβεβαιώσω και είναι σημαντικό να το πούμε ευθύ εξ αρχή. Εκτιμούμε ιδιαίτερω ε, τι εργασίε ε, του Ελληνικού Συνεδρίου έχει, των Ελληνικών. Έχει ε, εντοπίσει πολύ σωστά προβλήματα που υφίστανται στο πλαίσιο του EIT, προβλήματα ω προ τι πρακτικέ εργασιών, προ τον τρόπο αλληλεπίδραση με τα KICS, προβλήματα που ε, τους απέτρεψαν να επιτύχουν ε, τα αποτελέσματα που δεχόμενος θα ήθελαν. Αποδεχόμαστε πλήρως ε, τις συστάσεις που έχουν γίνει από το Ελληνικό Συνέδριο και σκοπός τώρα είναι να εξετάσουμε την υλοποίηση αυτών των συστάσεων. Συμφωνούμε απολύτω με την ανάλυση ότι το επιχειρησιακό πλαίσιο ε, έχει γίνει εξαιρετικά περίπλοκο, ότι η μέτρηση των επιδόσεων θα μπορούσε να είναι πιο σαφής. Ήδη εξετάζουμε και ως Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κινητοτομίας και Τεχνολογίας και τα ΚΙΚΣ για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολυετή ε, καθορισμό του προπολογισμού δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια, γιατί το ελεγκτικό συνέδριο υπό το πλαίσιο της συμμόρφωσης δεν θα ήθελε να κινηθούμε εξαιρετικά γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα και να μην λάβουμε υπόψη ε, τους ισχύοντες ε, κανόνες. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε ποιο είναι το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα, ενδεχομένως 2017, πιο πιθανό το 2018. Έχουμε όμως ξεκινήσει. Άλλα ζητήματα που ανέφερε ο κύριος Μπρένικ Μάιερ στην ε, παρουσίασή του. πώς θα δώσουμε μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία και ανεξαρτησία στα EITs. Ήταν εδώ και ο Ερμόδιος Επίτροπος είναι ορισμένες εβδομάδες στην Επιτροπή σας. Τώρα για την ενίσχυση του προσωπικού. Αυτό ανακύπτει ξανά και ξανά ε, τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα συνεχές πρόβλημα ε, στο EIT. Ε, και στα μέλη του προσωπικού και σε επίπεδο διοίκηση. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση του τελευταίου μήνε και το EIT μα λέει ότι θα συνεχίσει αυτή η βελτίωση. Για την ολοκλήρωση τη δομή του προσωπικού, αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και θα προταθούν και άλλε λύσει στο προσεχέ μέλλον. Η ομάδα υψηλού επίπεδου που έχει συστήσει ο κ. Ναύρατσιτ ήταν εδώ πριν μερικέ εβδομάδε, ε, Πρόεδρε. Ο Επίτροπο Ναύρατσιτ ανέφερε την πρόθεσή του σύσταση μια τέτοια ομάδα. Έχει αρχίσει τι εργασίε τη. Δεν θα επισέλθει τώρα στι τεχνικέ λεπτομέρειε ε, κάποιον από τα ζητήματα που ανέφερε η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Θα επικεντρωθεί στα βασικά ε, στρατηγικά ζητήματα που έχουν ε, αναφερθεί στην έκθεση, όπως η μεγάλη πρόκληση της επίτευξης της βιωσιμότητας ε, μακροπροθέσμους ε, του ΚΙΚΣ και του EIT, το οποίο αναγνωρίζεται ως μείζωνα πρόκληση. Και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν την ομάδα υψηλού επίπεδου. Μετά, επίσης θα την απασχολήσει η εντολή του EIT να αποτανθεί προς ε, υπερπροσωπούμενες περιφέρειες Υπάρχουν δυσκολίες λοιπόν σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη ορισμένων περιφερειών στο έργο. Γι' αυτό θα το εξετάσει με μεγάλη προσοχή και άλλα τέτοια μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. Πώ το ΙΑΤ θα ενταχθεί στο ευρύτερο οικοδόμημα τη Ευρωπαϊκή Πολιτική καινοτομία. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να απαντήσω σε ορισμένα από τα ερωτήματα και σχόλια που ανέφεραν τα μέλη. Ο κύριος Έλλερ έθεσε το ζήτημα το αν η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τώρα αντικατοπτρίζει τους αρχικούς κανόνες που θεσπίστηκαν δηλαδή εξ αρχής ε, ή κάποιε λανθασμένε πρακτικέ. Θα ήθελα ενδεχομένω και ο ίδιο ο διευθυντή να τα σχολιάσει, αλλά εγώ από πλευρά τη Επιτροπή να πω ότι είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Βλέπουμε λοιπόν, και αυτό σωστά αναφέρεται και στι συστάσει, ότι πρέπει να επανεξετάσουμε και τη νομική βάση. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν συνδέονται με την διεύρυνση ε, της νομικής βάσης του ΙΑΤ, e αλλά συνδέονται με την υποχρέωση να εξετάσουμε το μηχανισμό. Και αυτός είναι καλός στόχος. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να αποτελεί μοχλό ε, χρηματοδότησης από άλλους. Το θέμα όμω είναι πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Ίσως στη νομική βάση να προσδιορίζεται υπερβολικά. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αποδέχεται αυτό πλήρω. Εξετάζουμε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Ε, δεν ε, μας ενθουσιάζει η ιδέα της τροποποίησης της νομικής βάσης, όμως ενδεχομένως να χρειαστεί για να άρουμε ορισμένους φραγμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή γιατί μπορεί όντω να βελτιωθεί το εργασιακό περιβάλλον ε, του EIT. Ο κύριος Ρούμπικ μας επενθύμησε ότι το EIT ουσιαστικά είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο. Και είναι σημαντική αυτή η υπενθύμηση. Και στις συζητήσεις μας, ε, και εμείς είπαμε ότι είναι σαν να ξεχνούν ε, ε, την σημαντική συμβολή του EIT ε, στην εκπαίδευση. Μας έβλεπαν μόνο ως μοχλό καινοτομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα υπάρξουν σημαντικέ επιτυχίε ε, στο μέλλον, καθώ θα αποφυτούν και περισσότεροι φοιτητέ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Είναι λοιπόν σημαντική υπενθύμηση ότι βασική αποστολή του EIT ήταν να πάρει γνώσεις που παράγονται στις υποδομές και να τις συνδυάσει με την αγορά και τη βιομηχανία και, και τον κλάδο δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε έτσι να έχουμε ε, εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες και πολλή καινοτομία. Αυτός είναι ο στόχος που νομίζω ότι ευσταθεί. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε και θα εφαρμόσουμε και αυτές τις συστάσεις που αναφέρει η έκθεση. Τώρα, γιατί πρέπει να επαναξετάσουμε την νομική βάση. Νομίζω, όπως απάντησα και στον κύριο Έιλερ, να επαναξετάσουμε λοιπόν την νομική βάση, όχι για να τροποποιήσουμε εκ βάθρων ε, τον τρόπο αυτόν ε, συγκερασμού της ε, παιδείας και της αγοράς εργασίας και του κλάδου, αλλά πώς θα βρούμε ακριβώς ε, πρακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής βιωσιμότητας και το ζήτημα της ε, μη ευρωπαϊκής θεματοδότησης. Αυτά είναι τα θέματα που μας οδηγούν ε, στο συμπέρασμα ότι πρέπει όντως να επανεξετάσουμε την νομική βάση. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η δέσμευση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EIT είναι υπέρ μιας αναθεώρησης και πιστεύουμε ότι έτσι θα γίνει ε, το EIT ένα πιο ισχυρό μέσο για το μέλλον. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις εξηγήσεις σας και παρακαλώ τον κύριο Μπρένιγκ Μάιερ, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να μας δώσει κάποιες απαντήσεις από την πλευρά του θεσμικού σας οργάνου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά να απαντήσω για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Μάλλον για λόγου οικονομία, θα μην πάρα πολύ σύντομο, γιατί ο εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχολίασε κάποια πράγματα με τρόπο πάρα πολύ εύστοχο και ενημερωτικό. Στα γερμανικά, αξιότιμε κύριε Έλερ, θέσατε μια πολύ σημαντική ερώτηση. Και απαντώ στα αγγλικά. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια είναι η βάση τον παρατηρήσεών σας. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο. αιτία είναι 2008-2015. Τα πρώτα επτά χρόνια της λειτουργίας του Ινστιτούτου. Και στο τέλος έχουμε σταθμίσει όλες τις πληροφορίες και τι παρατηρήσαμε μετά από μια επταετή λειτουργία. Ότι κανονικά είναι αρκετό διάστημα για να δεις κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και είδαμε λοιπόν όντως ότι τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά. Θα έπρεπε να είχε προκύψει περισσότερη δουλειά. Μεγάλη γραφειοκρατία, μεγάλη δίκηση. Η προσέγγιση ήταν ιδιαίτερα γραφειοκρατική και βασιζόταν πάρα πολύ στη λογοδοσία και πολύ λίγο στην καινοτομία. Και ξέρετε, η καινοτομία από τη φύση της είναι εύθραυστη, διότι ε, καμιά φορά ε, είναι χρήσιμη και η αποτυχία. Στην καινοτομία πραγματικά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Πού καταλήξαμε λοιπόν, ότι είναι πολύ μικρό το αποτέλεσμα, θα μπορούσε να υπάρχει πολύ μεγαλύτερο και έρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Έλερ και της κυρίας Μούντι. Εσείς ε, προτείνατε το εξής. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί ή απλώς να βελτιωθούν οι επιδόσεις. Και απάντησε πρόσωπος της Ευρωπαϊκή Επιτροπής και το επαναλαμβάνω σύντομη, είναι και τα δύο. Και τα δύο. Υπάρχουν κάποια βασικά προβλήματα στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, οι συμπροματικές δραστηριότητες επειδή δεν εμφανίζονται θα πρέπει να τους αποκλείσουμε. Αλλά από την άλλη η αηφορία και η βιωσιμότητα των προγράμματων είναι πολύ σημαντική και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Άρα το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με το αν πάει κάτι στραβά διορθώστε το. Εν μέρη διορθώνεται αυτό και εν μέρη αναπτύσσεται περισσότερο ε, η λειτουργία βάσει των αποτελεσμάτων. Η μελέτη τι στόχο έχει. Να δώσει ένα feedback ε, για τη λειτουργία και να βρεθούν βελτιώσεις για το μέλλον. Αξιότιμε κύριε Ρούμπιχ, στα γερμανικά τώρα είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας, αλλά θα την απαντήσω στα αγγλικά. Για την επιστήμη και την τεχνολογία. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι συνήθως αυτά τα δύο και μάλιστα πολύ συχνά είναι χωριστά. Και γενικά το Ινστιτούτο καινοτομία και τα κέντρα γνώσης συνεισφέρουν ε, σε μια διεπιστημονική ε, προσέγγιση και θα πρέπει να μεταφερθεί αυτή η διεπιστημονική γνώση στον έξω κόσμο, στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη λειτουργία όλων αυτών των θεμάτων. Τελευταίο, το, χρονικό πλαίσιο, όλες οι συστάσεις συνοδεύονται από ένα πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και το ελέγχουμε όπως και εσείς ελέγχετε ως πρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Έλλερ θέλει να προσθέσει κάτι, ένα σχόλιο. Δεν είναι σχόλιο ερώτηση πραγματικά, παρόλο που έχω τάση να κάνω σχόλια. Για τη γεωγραφική ε, αναφορά που κάνατε, η ισορροπία. Τα περισσότερα και αυτή τη στιγμή είναι στη Γερμανία. Αλλά το πλαίσιο είναι ορίζον 2020 και η γεωγραφική ισορροπία ε, έχει σημασία. Αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει η αριστεία και λιγότερη η γεωγραφική ισορροπία. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την έλλειψη ισορροπίας. Τώρα έχει σημασία η γεωγραφική κατανομή ή, ή τίποτα άλλο. innovation, so the, the, the purpose. Ε, το θέμα είναι η καινοτομία που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν. Αυτό μας νοιάζει η αριστεία και οι επιδόσεις ή που θα βρίσκονται γεωγραφικά. Αν είναι τα πάντα στη Φιλανδία, αν η Φιλανδία είναι η καλύτερη για αυτό το τομέα, γιατί όχι γιατί ε, το EIT είναι τμήμα του ορίζοντα 2020 και ορίζοντα 2020 είναι ε, ένα από τα λίγα πράγματα που δεν παίζει ρόλο η γεωγραφική ισορροπία αλλά η αριστεία. Ε, μπορείτε λίγο να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εν συντομία και πάλι. Αφενός, πολύ σωστά αναφέρεται ότι ο ορίζον 2020 δεν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική ισορροπία. Από την άλλη όμως, βλέπουμε ότι η ανάπτυξη και εξέλιξη προς τη γνώση και η μετάφραση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ε, σε καινοτομία και συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, ερευνητικών Ινστιτούτων και επιχειρήσεων πρέπει να είναι αποτελεσματική. Γι' αυτό και η παρατήρηση του Ελληνικού Συνεδρίου είναι ότι θα πρέπει να διευρυνθεί. Γιατί η εικόνα που έχουμε προς την γεωγραφική ισορροπία είναι περιορισμένη. Ο κ. Πολ Στέφορτ, επικεφαλής της ε, ομάδας, παραπέμπει στη σελίδα 43 της εκθεσής μας, όπου αναφέρουμε ότι αν υπάρξει Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ή μάλλον ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται εάν έχουμε συγκέντρωση υποδομών και πόρων σε λίγες μόνο χώρες. Πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν, ελπίζω έτσι να σας απαντώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Περισσότερου εδώ σήμερα. Πάντα μας, ε, μας ε, ενδιαφέρουν τέτοιου είδους δραστηριότητε και πρωτοβουλίες και τομείς όπως ε, στα Ινστιτούτα Ευρωπαϊκής ε, Καινοτομίας και ελπίζω και στο μέλλον ε, να σημειωθεί πρόοδος και βελτίωση στα σημεία που αναφέρετε στην έκθεσή σας. Και οι να είναι σαφείς για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Είναι σημαντικό αυτό τα Ινστιτούτα δηλαδή να μπορούν να βελτιώνουν ορισμένε αδυναμίε που πάντα υπάρχουν σε τέτοιου είδου Ινστιτούτα. Όμω από πλευρά εκπαίδευση, για παράδειγμα, είναι θετικό γιατί δημιουργείται μια νέα εικόνα. Πάντα ξεχνάμε την εκπαίδευση. Μιλούμε για καινοτομία, για επιχειρηματικότητα, αλλά σε αυτό το τρίγωνο της γνώσης δεν πρέπει να ξεχνάμε το ρόλο της εκπαίδευσης. Πρέπει λοιπόν να στηρίζουμε τέτοιες ε, πρωτοβουλίες. Ναι, ήθελα μόνο να ενημερώσω τους αδέλφους και τον πρόεδρο και να ενημερώσω και το ελληνικό συνέδριο για μια πρόσκληση Ήδη υπάρχει στη μέσα διάταξη της μόνιμης ε, Επιτροπής ε, Ομάδας Εργασίας για τον Ορίζοντα. Νομίζω το Σεπτέμβριο αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα. Αν συμφωνείτε κι εσείς και αν ενδιαφέρονται και οι συνάδελφοι, παρακαλώ, ελάτε. Είναι ανοιχτές οι συναντήσεις, όχι μόνο για τα μέλη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, Ας περάσουμε στο τελευταίο σημείο της σημερινής διάταξης κατά τη διάρκεια της πρωινή συνεδρίασης Χωρίς καμία καθυστέρηση λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τι ε, αποζημιώσεις και οικονομική. Συγγνώμη, ευθύνη αποζημιώσεις και χρηματοοικονομική ασφάλεια για τις επεράκτητε δραστηριότητες εκμετάλλευσης και τα σβάτα μετρελαίου και φυσικού αερίου. Νίκολα Μπέι. Εισηγητή. Ε, θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. σε σχέση και με την οδηγία για την υπεράκτη ασφάλεια. Για την Επιτροπή μας, Επιτροπή Αρμόδια για αυτά τα ζητήματα, η οδηγία είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής Βιομηχανίας που με υποστήριξη ε, στην εκπόνηση της νομοδότησης για την ευθύνη, την αποζημίωση και ε, τις ε, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανοιχτή θάλασσα. Ε, ξέρετε ότι αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Γιούρι. Στις 4 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε αυτό. Λέει όμως η Ευρωπαϊκή Επιστροπή και παραθέτω, κανένα ε, ε, μεγάλο ατύχημα δεν είχαμε από το 1988 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατάφεραν να βγάλουν τα διδάγματα οι εταιρείε από το Piper Alpha, το τρομερό αυτό δυστύχημα. 73% του πετρελαίου και φυσικού αερίου που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από κράτη-μέλη που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα, ε, άρα έχουν ε, τις ε, πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Το σχέδιο γνωμοδότης Επιτροπής Περιβάλλοντος μόλις κατατέθηκε και θα συζητηθεί την άλλη Τρίτη και αναφέρει την καταστροφή του 2010 στον κόλπο του Μεξικού, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι το κοινό μας πλαίσιο έκτοτε έχει ενισχυθεί για να μην προκύψει παρόμοια καταστροφή στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την οδηγία του Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων αυτών σε ανοιχτή θάλασσα. Θα πρέπει να προσθέσουμε και το πρωτόκολλο offshore που ενέκρινε το Συμβούλιο της ε, Σύμβασης της Βαρκελόνης. Η δική μας απόφαση ελήφθη για να προληφθούν όσο γίνεται καλύτερα τέτοια ατυχήματα με ανταλλαγή πληροφοριών και σα παραπέμπω στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παραθέτει κατάλογο εκτενή αυτών αυτών των διατάξεων. Επίσης, ε, οι εταιρείε τα τελευταία χρόνια έχουν επενδύσει γενναία ε, σε νέα συστήματα ασφαλείας και ιδιαίτερα η τεχνολογία well well-capping, όπως ονομάζεται, δηλαδή πολύ γρήγορα ε, στο ίδιο, στην ίδια την γεώτρηση και την πετρελοπηγή κλείνουν την πετρελοπηγή όταν υπάρχουν διαρροές. Η οδηγία του 2013 θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά πριν να αρχίσουμε να ζητούμε νέες ε, ποινικέ ευθύνε ε, πέρα από τι αστικέ και τι περιβαλλοντικέ που είναι σήμερα δεδομένε. Το παράρτημα Α, με άλλα λόγια, τη οδηγία του 2014 για την περιβαλλοντική ευθύνη δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί για να συμπεριλάβει την οδηγία 2013. Σε περίπτωση δυστυχήματο, η οδηγία αυτή του 2013 προβλέπει ε, την ευθύνη. Την έχει εκείνος που έχει την άδεια ε, να προβαίνει σε τέτοιες δραστηριότητες. Άρα ε, εδώ καθιερώνει τη αρχή ο πληρώνει. Σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και, και πάλι σε περίπτωση ατυχημάτων, θυμίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ήδη και θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η ευελιξία έτσι ώστε κάθε εταιρεία και φορέας να μπορεί να επιλέγει το καλύτερο μέσο ανάλογα με τι συνθήκε που επικρατούν σε κάθε έργο. Όπω εχθέ θύμισε ο πρόεδρο Μπούζεκ, μετά την παρουσίαση τη δική του έκθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι εδώ διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα των ε, πετρελαϊκών ε, εταιριών και φυσικού αερίου και είναι οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών. Πρόκειται για ενεργειακό εφοδιασμό που θέλουμε να είναι και ασφαλής αλλά και προσιτός οικονομικά για τους πολίτες μας. Δεν θέλω λοιπόν να βάλουμε επιπλέον εμπόδια ε, στις εταιρείες που έτσι και αλλιώς πολύ συχνά ταλαιπωρούνται από πολύ βαριές διατάξεις που ισχύουν σε εμά και δεν ισχύουν για τους νης ανταγωνιστές. Στις πρακτικές λεπτομέρειες έρχομαι. Σε αντίθεση με όσα ακούσαμε την Τρίτη, μέχρι τις 31 Μαΐου έχετε προθεσμία για τροπολογίες, άρα μην ε, βιαστείτε. Ε, θα δώσω διάφορες ε, ημερομηνίες στους και ηγητές συναδέλφους για να μπορέσουμε να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Βεβαίως είμαι στη διάθεση του καθενός αν θέλετε να συζητήσετε και να υπερασπιστείτε ένα βασικό κλάδο που είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες και εταιρείε φυσικού αερίου είναι στον πυρήνα και την καρδιά των οικονομιών μας. Ευχαριστώ. Thank you very much, um, Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Εξ ονόματος του σκιώδη ηγητή του ΕΛΚ ε, θα διαβάσω εγώ το κείμενο Είναι ο κύριος Μπέντσεν, ο οποίος απουσιάζει και θα σας αναγνώσω τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης ή της ομιλίας που μου έχει δώσει για να τα πει. Δυστυχώ όμω καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίε και προβλήματα στι μετακινήσει από και προ τι Βρυξέλλε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα πριν τι 12 το μεσημέρι. Άρα η ΡΕΑ απουσιάζει και δυστυχώ. Σα διαβάζω αυτά που μου έδωσε ο κ. Μπένσεν. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την, ε, το σχέδιο έκθεση που γενικά βρίσκουμε ικανοποιητικό στο ΕΛΚΑ. Θέλουμε να στηρίξουμε την αποφυγή της υπερβολικής νομοθεσίας καθώς και τα διοικητικά βάρη σε ένα τομέα όπου οι διεθνείς συμβάσεις και οι συμφωνίες υπάρχουν ήδη. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ε, περαιτέρω ευρωπαϊκή εναρμόνιση σε αυτό το τομέα της ευθύνης και της αποζημίωσης μπορεί να χρειαστεί στο μέλλον. Ωστόσο, είναι σκόπιμο και στηρίζεται και από την υπεράκτη βιομηχανία καθώς και από άλλους βουλεκόμενους ε, φορείς να, να, να εφαρμοστεί η οδηγία περί ασφάλειας, υπεράκτης ασφάλειας. Μετά η Κομισιόν θα αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω δράση περαιτέρω ενέργειε. Η... Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η γνωμοδότηση ως ευκαιρία για να τονιστεί η σημασία της υπεράκτης βιομηχανίας που αυξάνεται διαρκώς, όχι μόνο για την ασφάλεια στην ενέργεια, αλλά και για την ευρωπαϊκή οικονομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν ήταν ολόκληρη η ομιλία, αλλά προσπάθησα να σας αναφέρω τα πιο σημαντικά τμήματα. Mr. Ενώ, γιατί ο κύριος Μπέντς είναι ο ισκιώδης συζητητής του ΕΛΚΑ. Σοσιαλιστές. Κυρία Μίρια Μντάλη, σκιώδης. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, των Σοσιαλιστών θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή και ε, έχει φανεί η αξία της θέσπισης μέτρων ασφαλείας πριν να συμβούν ε, μεγάλα ατυχήματα. Γνωρίζουμε ήδη πως τα κρατημέλη ήδη ε, έχουν καθεστώτα ε, για την υπεράκτη ασφάλεια. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε φυσικά αυτές τις βιομηχανίες, αλλά να εξασφαλίσουμε πως θα φέρουν την ευθύνη για κάθε ζημιά και απώλεια ε, λόγω ε, υπεράκτιων ατυχημάτων. Είμαστε πολύ περήφανοι για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου που συμβάλλει εξαιρετικά στην κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια, στην απασχόληση, όπως σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε, για την απασχόληση υψηλά εκπαιδευμένου προσωπικού από ολόκληρη την Ένωση, αλλά και επειδή συμβάλλουν στην έρευνα και την ανάπτυξη και φυσικά είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλειά μας ε, ανεφοδιασμού ενέργεια. Αν και η παραγωγή πατρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο αριθμός των υπερακτίων εγκαταστάσεων θα αυξηθεί στο μέλλον, μάλλον ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα. Και ταυτόχρονα ε, τα υπεράκτητα ατυχήματα έχουν ε, μεγάλες επιπτώσεις για την αλληλευτική βιομηχανία και για την τουριστική βιομηχανία, καθώς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά αυτές οι οποίες εξαρτώνται ιδιαίτερα ε, από τις συνθήκες του κοινού θαλασσίου περιβάλλοντος για να μπορέσουν να εργαστούν. Να θυμίσουμε ότι οι οικονομίες η οικονομία επλήγει στα τελευταία ατυχήματα λόγω του ε, των ε, ετοιμάτων αποζημίωσης ε, ε, αν ήρθε στα 96% θα πρέπει γι' αυτό λοιπόν να θεσπιστεί το κατάλληλο πλαίσιο ώστε να αποζημιώνονται οι αλληλείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλοι όσοι επηρεάζονται από τέτοιο είδους ατυχήματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν τριών ειδών ευθύνες, περιβαλλοντική, αστική και ποινική ευθύνη και ε, ενώ υπάρχει εναρμόνιση για την ευθύνη για περιβαλλοντική ζημιά, για τα διάφορα είδη οικονομικής απώλειας δεν υπάρχει εναρμόνιση στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική απώλεια που σχετίζεται άμεσα με ένα τύχημα. Όσον αφορά τώρα την ποινική ευθύνη θα ήταν μέγα βήμα, πιστεύουμε, αν κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά που οδηγεί σε ατυχήμα, υπεράκτη ατυχήματα χαρακτηριστεί και περιλευθεί στην νομοθεσία, και θα είναι ένα ακόμα στρώμα πέρα από την ε, αστική και την περιβαλλοντική ευθύνη και πιστεύουμε πως η Κομισιόν θα πρέπει να βρει ε, ε λύσεις όσον αφορά την έλλειψη ε, ασφάλειας ε, με μέσα οικονομική σταθερότητα. Θέλουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και χρειαζόμαστε περισσότερε εγγυήσεις από πλευρά τη Κομισιόν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ισχυρίζεται ότι είναι πολύ νωρί ώστε να αξιολογήσει σωστά αν το ποινικό δίκαιο τη Ένωση είναι, είναι απαραίτητο για να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα υπεράκτη ασφάλεια στην Ένωση. Θα πρέπει ε, καταρχά να έχουμε περισσότερη εμπειρία. Εμεί πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε να γίνει ένα μεγάλο ατύχημα. Θα πρέπει να εξετάσουμε το πλαίσιό μας και αν αυτό λειτουργεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ρήτρε ασφαλείας, τις δεκλίδες ασφαλείας, ώστε να μπορούμε ε, πρακτικά να εμποδίσουμε τα ατυχήματα στο μέλλον και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για τη δουλειά του καθώς και του σκιώδες. Ευχαριστώ Τάραντ που ε, αντικαθιστά την κυρία Ριβαζή και μιλά εξ ονόματος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Κύριε Βεζή και ενδεχομένω να μην. Ε, το Μισελ. Τη Μισελ Βεζή μου ζήτησε να την εκπροσωπήσω. Πριν από έξι χρόνια είχαμε ακριβώς αυτή την καταστροφή του, της Deepwater Horizon, όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι. Γι' αυτό και ιδίω σήμερα θα πρέπει να θέσουμε ένα ερωτηματικό δίπλα στο επιχείρημα ότι υπάρχει υπερβολική ρύθμιση του κλάδου. Αυτό που θα ζημίωνε πραγματικά την ανταγωνιστικότητα του κλάδου των, ε, του πετρελαίου θα ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα. Γι' αυτό και έχουμε και την οδηγία σήμερα που προσπαθεί να θέσει πρότυπα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω, ε, πολλά ζητήματα ακόμα παραμένουν στην εθνική αρμοδιότητα και δεν έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να δούμε κατά πόσο είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της οδηγίας. Σε πολλά κρατημέλη δεν υπάρχει, για παράδειγμα, ε, σιγουριά ότι όλοι οι εμπορευόμενοι έχουν ε, τις, ε, τα περιουσιακά στοιχεία για να αποζημιώσουν ε, τους πληγέντες από τέτοια ατυχήματα και ενδεχομένως να συμπληρωθούν από τα χρήματα φορολογουμένων. Η οδηγία σήμερα λαμβάνει υπόψη την αρχή ορυπαίνων πληρών, όπως αναφέρει και ο Όμω μόνο για περιβαλλοντικέ ζημίε όχι ε, για ζητήματα δημόσιας ευθύνης. Όμως, ε, μια πετρολοκυλίδα δεν επηρεάζει μόνο την βιοπικιλότητα, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα, την αλληλεία, την υδατοκαλλιέργεια, τον τουρισμό και το καθεξής. Μετά, όχι μόνο το άρθρο το 194 της Συνθήκης για της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφορά και το 192 και 191. Επομένως, θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε ε, τέτοιου είδους αδικήματα, ο, ιδίως εάν υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων και νομίζω ότι και στο τίποτα χωράζον συνέβη αυτό γιατί υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εμπορευμένων και αριθμιστικών αρχών. Γι' αυτό προτείνουμε ε, να γίνουν έλεγχοι ασφαλείας από τον Ευρωπαϊκό ε, Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και όχι τόσο από τις εθνικές ε, υπηρεσίες που κάποιες φορές δεν είναι ανεξάρτητες εξαιτίας ε, πολιτικών ε, λόγων και μονοπωλίων που υπάρχουν σε συγκεκριμένες χώρες. Αυτά ήθελε να μου αναφέρει η κυρία Ρεβαζή και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος, για τις παρατηρήσεις σας. Η κυρία Σακοράφα. Ε, ε, υποκαθιστά τον κύριο Σουλκιώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε αντικαθιστώ τον κύριο Σιλικιώτη, ο οποίος δηλώνει ότι η ευθύνη των εταιριών για ζημίες από υπεράκτια ατυχήματα κατά την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε με προσοχή. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας καθορίζει το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να διεξάγονται οι δραστηριότητες στους ωκεανούς και είναι σημαντικό να εφαρμόζεται από όλους. Πέραν όμως αυτού, χρειάζεται να δούμε και πώς επιτυγχάνεται η ασφάλεια και με επιμέρους πολιτικές. Για την ομάδα μας, προτεραιότητα είναι να προωθηθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις και να ενισχυθούν τα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όλων των υπεράκτιων εργασιών, ώστε να ενισχυθεί πραγματικά η ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος των λαών. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι απαραίτητο να υπάρξει αλληλεγγύη και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε με διαφάνεια και μέσω της ανταλλαγής των απαραίτητων πληροφοριών να ενισχύσουμε τα συστήματα ασφαλείας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προωθήσουμε μέτρα για ενίσχυση της πρόληψης, καθώς επίσης και να εξετάσουμε εναλλακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την βελτίωση της διαθεσιμότητας των μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας, αλλά και για την διασφάλιση του άμεσου και κατάλληλου χειρισμού των αξιώσεων αποζημίωσης. Μονάχα έτσι θα είμαστε έτοιμοι όταν διαφανεί η ανάγκη και δεν θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ελλειπή μέσα χρηματοοικονομική ασφάλειας. Στη βάση αυτή θα είναι και οι τροπολογίε που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει κάποιος άλλο να πάρει τον λόγο. Ένα λόγο. Όχι. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Κύριε Στέφαν Μόζερ. Πνευματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βούζεκ, αξιότιμα μέλη, για την έκθεση, αλλά και για όλα τα σχολιά σας. Ε, εν γέννη συμφωνούμε με τα ευρήματα τα, και τις της έκθεσης, της νομοδότησης της Επιτροπής Ήτρα, γιατί όντως δεν υπάρχει λόγος για επιπρόσθετη νομοθεσία. Θα πρέπει ε, σταδιακά να εξετάζουμε βήμα το βήμα την ανάλυση μας, γιατί ήδη υπάρχουν διατάξεις ε, για την οικονομική ευθύνη σε ό,τι αφορά την ε, αίτηση για διοδότηση και τα, τα κράτη-μέλη λαμβάνουν υπόψη τη νομική ευθύνη για να προκειμένου να αδειοδοτήσουν. Αυτό συμπεριλαμβάνει και την οικονομική ασφάλεια και τη δυνατότητα ε, κάλυψης ε, της νομικής ευθύνη που θα πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορούμε λοιπόν να σας ε, διαβεβαιώσουμε ότι τα κράτη-μέλη ελέγχουν ότι οι αιτούντε έχουν επαρκή περιουσιακά στοιχεία, οικονομικού πόρου, για να μπορέσουν να καλύψουν τέτοιε επίγουσε καταστάσει σε περίπτωση κρίσης. Και θα πρέπει να έχουν ε, και λειτουργικές ε, διαδικασίες για την επαρκή ε, διαχείριση τέτοιων αξιώσεων αποζημίωσης. Αυτή τη στιγμή η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσο κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει καταλήλως όλα τα τμήματα της οδηγίας και τα έχουν μεταφέρει επαρκώς στην Εθνική Νομοθεσία. Και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συμβαίνει, για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή το αργότερο το 2019, όπως προβλέπει η οδηγία για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει ε, την πείρα που έχουν αποκομίσει από την εφαρμογή της οδηγίας και μετά θα έχουμε μια συνολική επισκόπηση της κατάστασης, εξετάζοντας και τις προσπάθειες από τις αρχές και να βρούμε κατάλληλες ε, λύσεις και προτάσεις εάν θεωρήσουμε ότι απαιτούνται βελτιώσεις. Και σίγουρα σε αυτή την έκθεση θα καλύψουμε και ζητήματα νομικής ευθύνης και αποζημιώσεων και οικονομικής ασφάλειας. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, να αντιδράσουμε προβολικά. Αυτό θα ήταν η θέσπιση επιπλέον νομοθεσία. Πρέπει να προχωρήσουμε με αναλογικό τρόπο και να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά και αν ε, χρειάζομαστε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος εισηγητής, παρακαλώ, για να απαντήσει. Καταληκτικά σχόλια, δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ. Τους κύριους εισηγητές για τα διάφορα σχόλιά τους. Θέλω να θυμίσω κάτι σημαντικό κατά την άποψή μου, ότι οι εταιρείε που ασχολούνται με τις δραστηριότητε αυτές είναι οι πρώτες που δεν θέλουν να υπάρξει ατύχημα και ε, είναι πάρα πολύ δρακόντια τα μέτρα που παίρνουν για την ασφάλεια. Ε, θα ήταν πάρα πολύ ε, άστοχο να προσθέσουμε ακόμα πιο τρακόντια μέτρα γιατί θα είναι ευαίσθητες και έφτραυσες και εκτεθειμένες έτσι στην διεθνή ε, ανταγωνιστική κατάσταση και οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να έχουν ε, υπερβολικά υψηλές απαιτήσει ε, που δεν ισχύουν για άλλους και υπάρχουν και έμεσες ε, συνέπειες και έμεσες ε, ζημίες που προκαλούνται από ένα ατύχημα, αλλά αυτό είναι μια τέρμονη διαδικασία γιατί πάντα υπάρχουν δευτερογενείς και τριτογενείς έμεσες συνέπειες και πάει λέγοντας μέχρι πού δηλαδή θα αποζημιώνουν και δεν θα πρέπει να ε, φέρνουμε σε δύσκολη θέση ένα κλάδο που είναι πολύ ελπιδοφόρος πάρα πολύ υψηλής τεχνολογίας και ε, δεν θα πρέπει να τον εκθέτουμε εμείς σε περαιτέρω και επιπλέον κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα και όλους τους κοιόδης ευχαριστούμε για ε, την καλή δουλειά. Τροπολογίες λοιπόν, προθεσμία ε, 31η Μαΐου στις 12 το μεσημέρι ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ στην ε, καθήλυνα αρμόδια που είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα, αρκετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω δύο λόγια τώρα ως feedback από τη συνεδρίαση των συντονιστών εχθές ε, το απόγευμα. Μερικά σημεία πάρα πολύ σύντομα οι συντονιστές αποφάσισαν να ορίσουν ένα μέλος στη Συμβουλευτική Επιτροπή ENTSO-E για τους διαχειριστές δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Η απόφαση για το πρόσωπο θα ληφθεί εν ευθέτω χρόνο από τη διάσκεψη των Προέδρων καταρχάς. Προτάσεις μπορείτε να στείλετε στη Γραμματεία μέχρι τις 11 Μαΐου. Άλλο σημαντικό ζήτημα η ανάθεση εκθέσεων εφαρμογή που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον πιστεύουμε, αποφάσισαν οι συντονιστέ να εφαρμόσουν το σύστημα που ισχύει με πληστηριασμό, αλλά να δημιουργήσουν ε, ένα ξεχωριστό λογαριασμό ή προπολογισμό πόντων για τις εκθέσεις εφαρμογή και τις νομοδοτήσεις. Πολύ ενδιαφέρον αυτό για τα μέλη μα, οι εκθέσει τέτοιου τύπου. Επόμενο θέμα. Αποφάσισαν οι συντονιστέ να αναβάλουν τη δημόσια ακρόαση για την επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης που είχε προβλεφθεί για τις 23 Μαΐου του 2016 για να γίνει άλλη ακρόαση εκείνη τη μέρα για το λεγόμενο χειμερινό πακέτο ή τη δέσμη μέτρων για το φυσικό αέριο. Και αυτό πάρα πολύ σημαντική απόφαση των συντονιστών διότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Ε... Είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Επόμενο θέμα. Ενέκριναν οι συντονιστές το πρόγραμμα δημόσιας ακρόασης για την οδηγία 4.0 ε, στις 14 ε, Ιουνίου του 2016 θα γίνει αυτό και τέλος συμφωνήσαμε και συζητήσαμε για τις μελέτες ε, τις ημερίδες μελέτες και τα εργαστήρια. Οι επαναπομπές αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ και στι 3 αρχίζουμε τη δημόσια ακρόαση με θέμα ρόλου τη αποθήκευση ενέργεια στο μελλοντικό ενεργειακό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας περιμένουμε πίσω στις 3. Ευχαριστώ πολύ. Okay.